Το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει ένα πραγματικά πολιτικό πρόσωπο στο πλαίσιο της κρίσης αυτής. Εξού και η ερώτησή μου. Σε συνέχεια και των ερωτημάτων του κυρίου Ντανζόν, του Προέδρου. Χθες ακούσαμε κάποιες προτεραιότητες. Αυτές πώς θα μεταφραστούν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και να υλοποιήσει μία ξεκάθαρη στρατηγική ή μήπως απλά θα πρέπει να παρετηθούμε και να δεχθούμε ότι είμαστε απλοί προσκεκλημένοι κάποιων συναντήσεων που οργανώνται από άλλους. Συγκεκριμένα τώρα για την αποστολή. Η έννοια διαχείριση της κρίσης εγκρίθηκε και το όλο δόγμα αυτό στα τέλη Μαρτίου. Και φαίνεται ότι Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες μεταξύ κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν, πού υπάρχουν διαφορές να μου πείτε. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις απόψεων σε ό,τι αφορά ε, το κατά πόσον θα, θα υπάρξει επέμβαση χερσαία στη Λιβύη ή πώς ακριβώς θα ε, οριστεί η χρήση της βίας και πώς θα ρυθμιστεί. Θα ήθελα να έχω απαντήσεις σε αυτά. Ποια ουσιαστικά είναι η περίμετρος, ποιο είναι το περίγραμμα της όλης αποστολής αυτής στη Λιβύη. Μπούτι Κόφερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά με την αδειά σας. Και θα ήθελα κύριε Παπόφσκι, δεν σκοπεύω να είμαι πολύ ευγενής, γιατί με απογοητεύσατε. πέραν του ότι δεν είμαι σε θέση να αντιληφθώ ποιες είναι αυτές οι γραφειοκρατικές ε, δυσκολίες οι οποίες ε, επιβάλλουν να έχουμε δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη, χωριστά εσά και χωριστά τον κύριο Ιώτσο και γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μαζί σα συζήτηση. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Αν δεν μπορείτε ούτε σε μια ημερήσια διάταξη να, ε, να συνεργαστείτε, πώς θα καταφέρετε στο ΙΕΣ e μέσα να κάνετε δουλειά. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είπατε τίποτα ουσιαστικό για την επιχείρηση. Θα μπορούσατε να μην έχετε ανοίξει καν το στόμα σα. Γιατί δεν μπορέσατε χτε οι υπουργοί να συμφωνήσουν για το κόλοψη, παραδείγματι. Το καθεστώ παρατηρητού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε, δεν έχει ε, συμφωνηθεί. Γιατί, ποια ήταν τα προβλήματα. Και θα έλεγα επίση, να πάμε λίγο πιο μακριά, γιατί στην 1η Απριλίου αποφασίστηκε και συμφωνήθηκε το management crisis concept χωρίς να ενημερωθεί το κοινοβούλιο. Γιατί δεν ενημερώθηκε το κοινοβούλιο. Αυτό το ορίζει η συνθήκη τη Λισαβόνα, Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Και με ένα καθήκον μου εδώ ω Ευρωβουλευτή είναι να ασκώ την ε, τις ευθύνες μου και τι αρμοδιότητες μου και ως προς την εξωτερική πολιτική. Εσείς όμως πήρατε αποφάσεις και δεν μας ενημερώσετε καθόλου και καθόλου δεν μου αρέσει αυτό. Οι battle groups, επί παραδείγματι, οι ομάδε κρούσεω τελικά, τι αποφασίσατε. Είναι μέσα στην έννοια αυτή, στο concept, τι δεν είναι. Τα κράτη-μέλη, τα εμπλεκόμενα, κάτω χώρε, Γερμανία, Φινλανδία, Αυστρία, Λιθουανία, συμπράττουνε. Σουηδία. Θα μας δώσετε κάποιες ουσιαστικές πληροφορίες. η κατάσταση στη Μισράτα. Από ό,τι μαθαίνουμε είναι η χειρότερη κατάσταση προ τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πιο επικίνδυνη. Ε, υπάρχει κάποιο στόχος για τη Μισράτα. Έχει μπει μέσα στο σχεδιασμό αυτών. Υπάρχει κάτι το οποίο σκοπεύετε να κάνετε. Και όπως και ο Πρόεδρος έχω την ίδια θέση ως προς την κατάσταση σχετική με την εκεχηρία. Πότε και πώ Έχει κάποιο νόημα να καθόμαστε εδώ και να σα ακούμε πράγμα που θα έπρεπε να έχει κάποιο νόημα, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ του τα όργανα. Αλλά εάν έχει κάποιο νόημα να σας ακούμε, παρακαλώ να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ο κύριος Βαν Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπουτικόφερ. Αυτή είναι η φύση του προβλήματος. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το ερώτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ε, για ανθρωπιστική βοήθεια δεδομένης της κατάστασης ε, στη Λιβύη. Υπάρχει όμως και ένα ξεχωριστό ζήτημα, το θέμα της εμπλοκής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπό το έμβλημα της ΚΕΠΑ. Εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί όλες οι προσπάθειες που κάνετε αφορούν την προσπάθεια ε, να υπάρξει άδεια από τον ε, ΟΗΕ να μπορέσει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το έμβλημα της ΚΕΠΑ. Πριν από μία εβδομάδα προσπαθήσατε ε, να υπάρξει κάτι τέτοιο σε θαλάσσια παρέμβαση για τη διατήρηση του εμπάργου όπλων, αλλά τα κράτη-μέλη είπαν όχι και είπαν ότι αυτό δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαίω. Τώρα μιλάμε για αυτό το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και μάλιστα να γίνει αυτό στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είστε απελπισμένοι να έχετε μία ακόμη αποστολή η οποία θα ε, διεξαχθεί στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και σε έξι μήνες όταν θα έχουμε ξεχάσει όλη τη Λιβύη και θα κάνουμε ε, ενημέρωση για την ΚΕΠΑ θα μιλάτε για 20 ή 21 αποστολές ε, στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και όλα αυτά πραγματικά είναι νοησίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα Ηνωμένα Έθνη είπαν στις συνεδριάσεις ε, PSE ότι δεν ε, θέλουν ε, να συμμετέχει στην, ανθρωπιστική, στην ανθρωπιστική βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατιωτικό τρόπο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να το καταπολεμήσει αυτό και προσπαθεί να πείσει με... και πρέπει να πω ότι όλες οι διπλωματικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται να, πάρει μια... να προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει κάτι στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Για όνομα του Θεού, ας επικεντρωθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα σε πράγματα που είναι χρήσιμα και που μπορούν να συμπληρώσουν τι δραστηριότητε των άλλων ε, οργανισμών. Αν θέλουμε στρατιωτική δράση, υπάρχει και το ΝΑΤΟ. Α ξεχάσουμε όλε αυτέ τι ανοησίε. Ο ε, πρόεδρο Φαντρόμπα στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα είπε ότι χωρί την Ευρώπη, χωρί την παρέμβαση τη Ευρώπη, θα είχε γίνει λουτρό αίματο στη Βεγγάζη τι να σα πω, για μένα αυτά είναι ανοησίες και τίποτα άλλο. Ε, αν δεν υπήρχε η Βρετανία και η Γαλλία και η παρέμβασή του όντω, ναι, τότε θα υπήρχε λουτρό αίματο στη Βεγγάζη. Οπότε, α είμαστε ε, ρεαλιστές. Αυτή είναι η πραγματική μου δυσκολία που έχω με όλο αυτό το πρόβλημα τη ΚΕΠΑ. Πραγματικά είναι μη ρεαλιστικό. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε κάτι που ουσιαστικά δεν υφίσταται, κανένας δεν το θέλει, αλλά όλοι βάσει περιπτώσει κάπως ε, το αποδέχονται γιατί θεωρούν ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Δεν είναι τίποτε το επιπρόσθετο, δεν, έχει καμία, δεν σημαίνει τίποτα από άποψη επιπρόσθετων πόρων. Οπότε αφήστε τη στρατιωτική πλευρά σε, όσοι κάνουν, σε όσους κάνουν τα στρατιωτικά. Επικεντρωθείτε σε ζητήματα όπως είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι στο πλαίσιο αυτό ε, μέσω της ΕΚΟ στην... Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την προσφορά ε, ανθρωπιστικής βοήθειας υπό τις συνθήκες αυτές και δεν χρειάζεται να γίνει αυτό στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Επίσης υπόθηκε ότι ο ΙΕ θέλει να μην τεθεί ένα αμφιβόλο η ουδετερότητά του ε, επουδενή. Ε, και γι' αυτό δεν θέλει τόσο την στρατιωτική παρέμβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει Εντάξει, ας μην πέφτουμε μόνοι μας σε κάποιο λάκκο που θα έχουμε σκάψει οι ίδιοι. Ας παρέχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, ας ξεχάσουμε την ΚΕΠΑ και ο κύριος Μπούντιγκόφερ ε, έχει τέτοιου είδους ανησυχίες οι οποίες έτσι θα επιλύονταν, όπως και ανησυχίες πολλών άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόσινγκ. Δεν μου τυχαίνει συχνά να συμφωνώ με τον κύριο Εν πάση περιπτώσει, η ιδέα να αφήσουμε την ε, στρατιωτική διάσταση και να επικεντρωθούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια μόνο με ικανοποιεί πολύ. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, κύριος Φανόρδον δυστυχώς δεν ακούγεται. Να συνεχίσω, λέει η κυρία Λεσί. Ε, γνωρίστε λοιπόν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ως προς την ε, U4 να συνεργαστεί με τις ε, δυνάμεις που έχουν οριστεί από το 2007 και ε, θα υπάρχει έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτής. Και επίσης, όπως είπε και ο κύριος Δονζόν, η ανθρωπιστική βοήθεια θα έχει σαν στόχο και την αλλαγή καθεστώτος. Επισημαίνω εδώ ότι για μένα ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια μόνο μετά από μια εκεχηρία μπορεί να υπάρξει. Αλλαγή προτεραιοτήτων θα σήμαινε ίσως και εξέλιξη ε, ως προς τη, ή μάλλον, ναι, ως προς τη θεώρηση των κινήτρων της ανθρωπιστικής βοήθειας. Λέτε επίσης ότι αποκλείονται οι δυνάμεις κατοχής. Εκπρόσωπος όμως του Υπουργείου Αμήνης Γερμανίας είπε ότι στη U4 θα μπορούσε να ανατεθεί και η ανάπτυξη δυνάμεων εδάφους, χερσαίων δυνάμεων. Αυτό έχει συγκεκριμένα προγραμματιστεί. Και αν ναι, δεν ισοδυναμώνει οι χερσαίες δυνάμεις με δυνάμεις κατοχής. Έχω ακόμα πέντε ε, συναδέλφους που στείλουν το λόγο. Θα σας παρακαλέσω να είμαστε σύντομοι όλοι για να προχωρήσουμε. Ο κύριος Λίσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάπως ε, παράδοξη αυτή η κατάσταση στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών. Ψηφίσαμε την έκθεση Κολκιέρη Εγώ ήμουν συντάκτης γνωμοδότησης για την έκθεση αυτή. Και εντωμεταξύ έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως ε, εξελίσσεται. Και αυτά που αναφέρονται στην έκθεση τελικά δεν ε, ακολουθούν ε, τις εξελίξει πραγματικότητας. Το σημαίνει ότι χάσαμε πολύ χρόνο και θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση προς τον κύριο Ποπόφσκι στην αρχή της παρέμβασής σας αναφερθήκατε στο ζήτημα της συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποιο επίπεδο λαμβάνει η χώρα αυτή η συνεργασία και θα ήθελα επίσης να ξέρω αν υπάρχει, μια, αν υπάρχει συνεργασία σε σχέση με τον προγραμματισμό για το όραμα για το μέλλον, δηλαδή για τα διάφορα σενάρια εξέλιξης της κατάστασης. Υπάρχει συνεργασία με ε, το ΝΑΤΟ και τα μέλη του ΝΑΤΟ και κυρίως αυτά που από στρατηγικής απόψεως είναι τα πιο ανεπτυγμένα. Ο κύριος Παλαιατσκής. Ε, ε, Ευχαριστώ. Από δική μου πλευρά, ένα ερώτημα. Εάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε στη διάθεσή μας κάποια αριθμητικά στοιχεία για το πώς αντιδρούν οι κοινωνίες μας, ε, οι κοινωνίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όσα συμβαίνουν στη Λιβύη, για την αντίδραση των μεγάλων χωρών, ε, του ΝΑΤΟ κτλ. Δηλαδή, τελικά η κοινωνία, η κοινή γνώμη είναι υπέρ ή κατά των δράσεων που αναλαμβάνουμε στη Λιβύη. Επόμενο ερώτημα. Η Ρωσία, η Κίνα, τι ρόλο έχουν. Υπάρχει συνεργασία με τις χώρες αυτές στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης στη Λιβύη από πλευράς μας. Ευχαριστώ. Κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ξέρω αν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν είχε προηγηθεί η, παρέμβαση του κυρίου Βανόρντεν. Η αλήθεια είναι ότι στην αντιμετώπιση της κρίσης της Λιβύης η Ευρώπη καθυστέρησε, εμφάνισε τα γνωστά σημάδια έλλειψη συντονισμού και αποφασιστικότητας που και στο παρελθόν έχει δείξει. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να θεραπευθεί αποτελεσματικά και το ταχύτερο δυνατόν. Και αυτό μπορεί να γίνει με την καλύτερη αξιοποίηση των προβλέψεων της συνθήκης τη Σαββόνα. Και χρειάζεται βεβαίως πολιτική βούληση. Αυτό είναι ένα. Υπάρχει λοιπόν έδαφος για να ασκηθεί κριτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προεκτείνουμε αυτή την λογική για την κριτική σε σημείο του να αγνοήσουμε ή να υποβαθμίσουμε πλήρως την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα εδώ, σαν αντεπιχείρημα στα όσα ακούστηκαν από τον κύριο Βανόρντεν, να θυμίσω σε όλους ότι για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος ασφάλειας είτε αυτό αφορά το διεθνές εμπόριο, είτε την ενέργεια, είτε ακόμα και την περιφερειακή ασφάλεια που είναι το πρόβλημα της πειρατείας στην περιοχή της Ομαλίας, ήταν πρώτη η Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε την επιχείρηση Ατλάντα με σημαντική επιτυχία και αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον ΝΑΤΟ και να κάνει μετά από καιρό μια παρόμοια επιχείρηση η οποία δεν ήταν και το ίδιο αποτελεσματική όσο εκείνη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να, το ε, κατηγορούμε συλλήβδιν και ουσιαστικά να αγνοούμε και να πετάμε στα σκουπίδια την προσπάθεια της Ένωσης να έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα ασφάλειας και άμυνας νομίζω ότι είναι μια λάθος προσέγγιση. Και εν πάση περιπτώσει βεβαίως έχουμε αδυναμίες αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά που πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Ο Τσόρτσιλ και επειδή μιλάω ως απάντηση στον κύριο Βανόρντεν, ο Τσόρτσιλ στον πόλεμο όταν ανέλαβε είπε «Μπορεί να μην είμαι λιοντάρι, αλλά σε μέναν έτυχε να πρέπει να βρυχηθώ» Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με την Ευρώπη. Μπορεί να μην είμαστε ακόμα λιοντάρια, αλλά έχουμε τον ρόλο και την πίεση και πρέπει να μπορούμε να βρεχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Madame eh, Presidente. Eu eh, tenho alguma dificuldade em compreender Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκοπό να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Λιβύη στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Κάτι το οποίο μπορεί να μην ε, ε, γίνει τελικά. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει αίτημα από πλευράς ε, ε, ΟΗΕ και του ΟΤΣΑ, του Γραφείου για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, οπότε δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει και αναρωτιόμαστε μήπως η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάτι συγκεκριμένο επιτόπου, εντάξει ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα στην περιοχή, την ευρύτερη, στη Σομαλία ή στις διάφορες γειτονικές χώρες, είναι ένα πραγματικό ερώτημα όμως αυτό του τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πέραν από τη δυνατότητα αντίδρασης, ανταπόκριση, υπάρχει βέβαια και το θέμα του νομικού πλαισίου, της νομικής βάσης. Έχουμε τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε το θέμα της προστασίας των αμάχων, αυτό φυσικά αποτελεί προτεραιότητα. Μπορεί να αποτελέσει αυτό λοιπόν μια στέρεη βάση για, την, ε, για μια, μια τέτοιου είδου παρέμβαση στο πλαίσιο τη ΚΕΠΑ, αλλά αυτά είναι τα όρια. Πέρα από αυτά τα όρια δεν υπάρχει κανένα αίτημα. Υπάρχει η απόφαση της 10ης Μαρτίου η οποία δεν θα είχε νόημα να εξελιχθεί σε μία οποιαδήποτε δράση στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ, για παράδειγμα, οποιαδήποτε παροχή εξοπλισμού ή οτιδήποτε τέτοιο. Είδατε τις ε, αποφάσεις του Βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οπότε, αντιθέτως με αυτά που είπε ο κύριος Βανόρντεν, εγώ πιστεύω ότι έχασε μια λαμπρή ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταστεί ορατή όσον αφορά το θέμα της ε, ε, πολιτικής, ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Και νομίζω ότι αυτή την ευκαιρία δεν την αξιοποίησε. Δεν συμφωνώ με όλα τα επιχειρήματα που μας παραθέσατε. Εγώ διαφωνώ με όλα αυτά τα επιχειρήματα, αλλά και με τα επιχειρήματα που ανέφερε η κυρία Άστον. Εντάξει, ακούγεται ότι τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν, ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συνένεση. Εντάξει, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά δεν υπήρξε και πρωτοβουλία από πλευρά ε, Άστων ε, τουλάχιστον για να μπορέσουμε να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε με κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ενώ στο πλαίσιο τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα θα ήταν ενδεχομένω δυνατό να γίνει κάτι στο πλαίσιο τη ΚΕΠΑ. Πρέπει όμω να υπάρχει μια πρωτοβουλία. Η βάση πρέπει να είναι μια πρωτοβουλία. Και τότε ναι, να διαφωνήσουμε. Αλλά δεν ρώτησε κανείς τα κράτη-μέλη αν συμφωνούν ή διαφωνούν με οτιδήποτε. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι θλιβερό. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες εξηγήσει από τον κύριο Ποπόφσκι. Μιλήσαμε όντως για εξοπλισμό των εξεγερθέντων, συζητήθηκε όντω το θέμα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ. Εγώ θα ήθελα συγκεκριμένε απαντήσει και θα ήθελα να ξέρω επίση αν συζητήσατε καθόλου ε, για την πρωτοβουλία που ε, ανέλαβε η Αφρικανική Ένωση. Συζητήσατε για το θέμα αυτό. Υπάρχουν και διάφορα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι η αποχώρηση από την εξουσία του Καντάφη ε, και να επιληφθεί του θέματος η, τη διεθνής δικαιοσύνη. Ε, συζητήσατε όλα αυτά τα θέματα, όλα, όλα αυτά τα, ε, θέματα που έθεσε η Αφρικανική Ένωση. Και Όσον αφορά τη δική σα θεώρηση των πραγμάτων, πώς βλέπετε τις εξελίξεις ε, σε σχέση, για παράδειγμα, με την αναδιάρθρωση ε, του ε, τομέα της ασφάλειας σε περίπτωση που παραμείνει ο, ο Καντάφη στην εξουσία. Κυρία Κοπά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ποπόφσκι, Τελώ υπό κάποια σύγχυση. Ε, έχουμε για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας την κατάσταση στη Λιβύη, χωρί όμως για μια ακόμη φορά να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Το δικό μου ερώτημα είναι ποιο είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιχείρηση. Αλλαγή του καθεστώτος, ε, ε, να φύγει ο Καντάφη, ε, υπάρχει κάποια σύγχυση, κάποια βεβαιότητα που μπορεί από επιχειρησική πλευρά να αποβεί και επιζήμια. Επί το που φαίνεται η κατάσταση να είναι τέτοια που κανένα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Γιατί η πολίτευση μέχρι τώρα δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει ε, την παρέμβαση τη Δύση και να υποφεληθεί από αυτήν και από την άλλη υπάρχει σημαντικός ε, κίνδυνος να παραταθεί διαμακρών αυτή η αντιπαράθεση και να έχουμε τελικά ένα αποτυχημένο ένα κράτος το οποίο θα καταρρεύσει. Το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Στις υπηρεσίες σας, στα σενάρια αυτά τα συζητάτε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι της ε, ΕΙΕΔ σε αυτή την ε, αντιπαράσταση, αυτή τη σύγκρουση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις, ε, πολλές παρεμβάσεις. Ο κύριος Ποπόφσκι για 10 λεπτά τουλάχιστον έχετε το λόγο. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Θα κάνω ό,τι μπορώ πάντως για να απαντήσω και θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις για να έχουμε έτσι κάποια δομή. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του, της κυρίας Γκόμης στην ερώτηση, είναι παρονοή, αλλά όχι παντού. Πράγματι, έχουμε και εμείς παρουσία επιτόπου, έχουμε την ε, γάμα δέλτα ΕΚΟ και παρουσία ε, του ΟΗΕ στη Μισράτα, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, δεν υπάρχει. Άρα όλοι βασιζόμαστε στις διαθέσιμες πηγές και αυτό περιλαμβάνει και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται με τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως είναι οι γιατροί χωρίς σύνορα ή ο Κάποια κράτη ε, με ζήτησαν, ε, για, μάλλον κάποιοι βουλευτές ρώτησαν για τα battle groups, τις μάχημες ομάδες. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο και δεν ξέρουμε ακριβώς τις ανάγκες. Ίσως χρειαστούν ε, κάποιες δυνάμεις εξειδικευμένες ε, θεωρητικά, αλλά δεν έχουμε εξετάσει ακόμη το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε μάχημη ομάδα. Γιατί είμαστε στο πρώτο στάδιο ακόμα που κάνουμε κάποια χαρτογράφηση της κατάστασης και των αναγκών που έχουν εντοπίσει ε, που θα εντοπίσει μάλλον ο διοικητή σε επιχείρηση που δεν το έχει κάνει ακόμη. Και θα ακολουθήσει η επόμενη φάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τον Γκαντάφη, χθε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ήταν κατηγορηματικό το Συμβούλιο λέγοντα ότι πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία και το αξίωμά του Καντάφη. Αυτό είναι σαφέ. Και γι' αυτό το σχέδιο δράση, αν θέλει το δικό χάρτη Αφρικανική Ένωση, δεν έχει γίνει αποδεκτός ανεφόρον από το Εθνικό Συμβούλιο στη Βεγγάζη γιατί το προσωρινό συμβούλιο λέει ότι πρέπει να φύγει άμεσα ο Καντάφη. Δεν θέλει να έχει καμία διαπραγμάτευση μαζί του. Ο Υπουργό Εξωτερικών ή οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν μια συζήτηση με τον κύριο Τσιμπρίλ που είναι ο εκπρόσωπος ε, του προσωρινού αυτού συμβουλίου. Έγινε χθε στο Λουξεμβούργο αυτή η ε, συζήτηση και ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες γιατί έγινε και κλεισμένο των θυρών. Ήταν ε, μια συνάντηση στην οποία εγώ προσωπικά δεν παριστα... Τώρα μπορεί κανείς να εκφράσει τις εικασίες του και τις υποθέσεις του για τα διάφορα σενάρια. Νομίζω ότι είναι σαφές και από τις σημερινές συζητήσεις στο Συμβούλιο μεταξύ άλλων ότι σίγουρα θέλουμε τη διχοτόμηση της χώρας να την αποφύγουμε. Είναι προφανές αυτό, αλλά αυτή η σύγκρουση αν παραταθεί, αν επιμηκυνθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να προβλέψει που θα οδηγήσει και ποια κατάληξη θα έχει όλη η κατάσταση. Και το θέμα ε, τη συμμετοχή των χωρών που θα ε, συμμετάσχουν στον συναφισμό συζητήσει σήμερα. Αυτό το, το καταλαβαίνω και το παρακολουθούμε. Εξετάζουμε τα διάφορα σενάρια, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στην ε, διάρκεια της εβδομάδας λίγο αργότερα θα προσπαθήσουμε να, έχουμε μια, να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης ε, αφού θα, έχει, ε, θα έχουν τερματιστεί ε, οι συγκρούσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, ακούστε, αυτό συζητήθηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα και γνωρίζετε ότι είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Διαφέρουν οι απόψει των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη, την εφαρμογή τη αρχή αυτή μεταξύ κρατών μελών και επειδή δεν εμπίπτει δική μου αρμοδιότητα, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο από αυτού. Πάντω, υπάρχει σχετική συζήτηση, η οποία γίνεται στα κατάλληλα βήματα συζήτηση. Και έρχομαι τώρα στη Frontex. Δεν ζήτησε κάποια ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέτρα δηλαδή και πά, άρα ίσως να μην χρειαστεί. Η εντολή άλλωστε της Frontex είναι ξεκάθαρη σε σχέση με το θέμα αυτό. Τώρα, μπορεί να μην απαντάω στη σειρά, ο κύριος Βανόρντεν τα είπε πολύ έτσι ξεκάθαρα για την ε, ΚΕΠΑ. Δεν θέλω να επισέλθω σε συζήτηση για την ΚΕΠΑ εμείς κάνουμε το σχεδιασμό μας. Έχουμε κάποιες, ε, κάποιες, κάποια όρια τα οποία μας τα απαγορεύουν τα κράτη-μέλη. Έχουμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και δεν πάμε πιο πέρα από όσο είναι έτοιμα να πάνε τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των επιχειρήσεων και πά. Τα κράτη-μέλη το συζήτησαν, κύριε Βανόρντεν. Κάποια κράτη-μέλη ήθελαν να εξετάσει το ενδεχόμενο της επιβολής εμπάργου όπλων ε, αλλά δεν ε, υπήρξε συμφωνία. Άρα έχει κάποιο νόημα να επιμείνουμε εμεί σε κάτι που βλέπουμε ότι δεν είναι έτοιμα να κάνουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό επικεντρωθήκαμε μόνο στο ανθρωπιστικό ζήτημα. Ούτε πιέζουμε το γραφείο του Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, το ΟΤΣΑ. Έκανε κάποια, είχε κάποια επαφή η κυρία Έμις με την κυρία Άστον. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποια αιτήματα, είτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε προς το ΝΑΤΟ, για ανθρωπιστική παρέμβαση, δεν αποκλείεται. Ε, είναι βέβαια μια τελευταία ε, λύση, ενδεχομένως θα είναι η τελευταία επιλογή. Δεν έχει ζητηθεί ακόμα, ίσως ζητηθεί. Κάποια σχόλια εκτός μικροφώνου. Σας παρακαλώ, ας αφήσουμε τον κύριο Παπόφσκι να απαντήσει, γιατί νομίζω ότι όλοι είχαν το χρόνο τους και μπόρεσαν να εκφράσουν τις γνωστές άλλωστε απόψεις τους. Κύριος Παπόφσκι, είναι εθνική η πόρια, έτσι, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι τα πράγματα. Θα επανέλθω και σχέση μας με τον ΝΑΤΟ. Ε, υπάρχει συμφωνία πάντως να μην δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου θα υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ για του ε, τους πόρους και μιλάω για τους στρατιωτικούς πόρους. Θα δούμε ε, τι θα γίνει αν χρειαστεί να εμπλακούμε εμείς προσωπικά ε, ως Ένωση. Τώρα, αποφασίστηκε να βάλουμε κάποια πλαίσια και να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι και σε σύντομο χρονικό διάστημα αν υπάρξει σχετικό έτοιμο από τον Ότσα, το Ότσα να παρέμβουμε. Τώρα, Κύριε Μπιτεκόφερ, είσαστε κάπως σκληρός απέναντί μου, αλλά δεν σας κρατώ κακία. Είναι νομίζω απαραίτητο να συναντιόμαστε μέσα στι ε, συνεδρίε αυτέ των επιτροπών, να ανταλλάσσουμε απόψει. Εγώ πάντα είμαι στη θέση σα και οι άλλοι συνάδελφοι ασφαλώ, όποτε θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο κάτι τέτοιο. Για τι battle groups, εν μέρει έχω απαντήσει πιστεύω, περισσότερα δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Τι είδου δυνατότητε θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, θα χρειαστούμε μάλλον να χρησιμοποιήσουμε στην ε, περιοχή. Δεν μπορώ να πω. Η Μιστράτα είναι μία περίπτωση είναι δηλαδή μια περιοχή όπου θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε δράση και αυτό πάλι θα προκύψει από τον περαιτέρω σχεδιασμό. Θα ληφθεί υπόψη ασφαλώς η κατάσταση. Και μια και άρχισα στα γερμανικά, συνεχίσω. Η κυρία Λόσινγκ μίλησε για το 2011 και τη Frontex. Η Frontex δεν έχει επιδείξει κάποια ανάγκη για ανάπτυξη δράσης ε, με υποστήριξη από μέσα της ε, ΚΕΠΑ. Όντως αποκλείονται δυνάμεις κατοχής, αυτό είναι σαφές και από το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αποκλείεται συγκεκριμένες δυνατότητες να αναπτυχθούν επί εδάφους, να χρειαστεί να εγκατασταθούν δηλαδή κάποιες δυνάμεις ε, του εδάφους είτε της Αιγύπτου είτε της Τινησίας και γι' αυτό ανέφερα τα κράτη αυτά ότι έχουμε επαφές μαζί τους και θα δούμε αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε να συμφωνήσουν, να μας επιτρέψουν στην επιχείρηση αυτή, να μας προσφέρουν υποστήριξη στην επιχείρηση αυτή. Πάντως δεν είναι δυνάμεις κατοχής αυτές οι χερσαίες δυνάμεις που θα χρειαστεί ενδεχομένως να επέμβουν σε μια τέτοια περίπτωση. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στη μητρική μου γλώσσα για να μιλήσω για τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ η οποία πηγαίνει καλά, προχωρεί καλά. Η κυρία Άστον είχε την ευκαιρία να προχωρήσει μια ανταλλαγή απόψε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα και επίσης να συζητήσει την κατάσταση των προετοιμασιών των δικών μας και της επιχείρησης του ΝΑΤΟ. Δηλαδή συζητήθηκε το τι είδους μέσα μπορούμε να έχουμε στη θέση μας. Όπως είπαμε πρόκειται για εθνικούς πόρους. Επίσης, όπως είπα, υπάρχει στενή συνεργασία Υπάρχει γραφείο συνδέσμου μεταξύ του δικού μας, ε, της δικής μας αρχής και της, ε, του Γενικού Επιτελείου του ΝΑΤΟ. Η κυρία στον Πέμπτη και Παρασκευή είναι στο Βερολίνο, σε συνάντηση του ΝΑΤΟ. με θέμα την κατάσταση στη Λιβύη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δημοσκοπήσεις στη Λιβύη. Δεν ε, διάβασα τίποτε στο Ευρωβαρόμετρο σχετικά. Με τη Ρωσία και την Κίνα ήρθαμε σε επαφή, αλλά κυρίως ε, στο πλαίσιο των ε, συζητήσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στις σχετικές συζητήσεις μόνο μιλήσαμε με τη Ρωσία και την Κίνα. Η ύπατη εκπρόσωπος ε, θα συναντήσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας κατά τις ερχόμενες ημέρες και φυσικά η Λιβύη θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Τώρα το ερώτημα του εξοπλισμού των ε, ε, εξεγερθέντων. Δεν υπάρχει συνένεση επί του θέματος αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εμπάργκο ισχύει και το εμπάργκο δεν είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν λέει ότι μπορούμε στο ένα μέρος της, ε, ε, στο ένα της, ε, της πολεμικής σύραξης να πούμε ναι και στο άλλο όχι. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο θα, θα υπάρξει μία βάση για να προοδεύσουμε στο Κάιρο, το, στην, στη συνάντηση που θα έχουμε αύριο των τεσσάρων οργανισμών. Και όσον αφορά τώρα την αναδιάρθρωση του τομέα ασφαλείας, οι εμπειρογνώμονές μας αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αναπτύξουν διάφορα σενάρια ενδεχόμενης εμπλοκής ε, στην ε, ε, περίοδο μετά την ε, μετά τις συγκρούσεις. Έχουμε κάποιες εμπειρίες ε, από τα Βαλκάνια, από τη Μέση Ανατολή, από το Κονγκό και θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες αυτές. Είναι γεγονός ότι η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΚΕΠΑ ε, για την προστασία των αμάχων και την αναδιάρθρωση μετά από τις συγκρούσεις ενδεχομένως ε, να συζητηθεί. Αλλά όλα αυτά αφού ολοκληρωθεί ε, αφού τελειώσουν οι συγκρούσεις. Όσον αφορά τώρα τον Καντάφη, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής ότι πρέπει να αποχωρήσει. Τώρα, οι αποφάσεις ε, από τον ίδιο το λιβικό λαό θα ε, παρθούν όσον αφορά το μέλλον της Λιβύης. Βέβαια αυτό υποθέτει και την αναγνώριση του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου που ε, έχει αναγνωριστεί ως συνομιλητής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών συνάντησαν τον κύριο Τζμπίλε χτες στο Λουξεμβούργο. Δεν θέλω να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση τώρα. Έχουμε πολύ περιορισμένο διάστημα στη διαθέσή μας. Μα δεν απαντήσατε στον κύριο Μπιτικόφερ στην ερώτηση για την παράξενη αυτή αλλαγή στον προγραμματισμό στην ημερήσια διάταξη. Το σημειώνουμε. Και βλέπουμε ότι δεν είναι από ό,τι φαίνεται διατεθειμένη η ότι θα ήταν καλό μάλλον να μην είναι διατεθειμένη η ΑΕΔ να ζητήσει χωδιαχωρισμό της μερισσίας διάταξης από τους άλλους προσκεκλημένους, όπως έγινε στη δική μας. Κύριος Μπιουτικόφερ. Δυστυχώς κύριε Παπόφσκι. Δεν με διαφωτίσατε. Σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ίδια από ό,τι φαίνεται διχαστική σχέση με τη Λιβύα όπως ο Ομπάμα, ο οποίος ως πολιτικός λέει ότι θα πρέπει να αποχωρήσει από την ε, θα πρέπει μάλλον να βοηθήσει στη διάσωση της Λιβύης, ενώ στρατιωτικός λέει ότι θα πρέπει να εμπλακεί ως επικεφαλής του στρατού. Το ενδιαφέρον ότι έχει πάθει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως. Δεύτερον, το να μου λέτε ότι η Μισράτα είναι πιθανός στόχος τι είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε, το ξέρω και μόνος μου, δεν σας ρώτησα αυτό. Δεν μου απαντήσατε όμως την ερώτηση στο πόσο σοβαρά παίρνετε υπόψη αυτή την κατάσταση. Δεν είστε βέβαιε αν θα χρησιμοποιήσουμε battle groups ή κάτι άλλο. Εάν πρόκειται να αναπτύξουμε battle groups, και βλέπω εδώ ένα έγγραφο του Συμβουλίου, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση ότι θα ε, το πράξουμε αυτό και μέχρι την εκκίνηση αυτής της αποστολής περνάνε δέκα μέρες. 10 μέρες που θα περάσουν τι θα γίνει στη Μισράτα. Και αν δεν πρόκειται να αναπτύξουμε battle groups, εβδομάδες και μήνε θα περάσουν πριν αναλάβουμε κάποια δράση. Μα λέτε λοιπόν ότι είναι πιθανό στόχο μιας δράσης Μισράτα και κατά τα άλλα δεν ξέρετε τι πρόκειται να γίνει. Περί του σύγχυση πρόκειται. Εάν πρόκειται να αναλάβουμε δράση πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα και Άρα να αναπτύξουμε battle groups και γρήγορα. Διαφορετικά το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και παρακαλώ να σταματήσετε αυτές τις, ε, αυτές τις δίθεν ε, ενημερώσεις, γιατί αν νομίζετε ότι μας ε, ικανοποιούν και ότι μας πείθετε, απατάστε. Και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το εξή από το computer, από το Spiegel Online, το περιοδικό, που λέει, παραθέτω, από ό,τι μας είπε ένας ε, στρατηγός, ξεκίνησε την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων το ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και την στρατιωτική διασφάλιση της κατάστασης στην Λιβύη, από ό,τι είπε ο κύριος Μάνφριτ Λαμπ ε, σε μια συνέντευξη σε γερμανική τηλεόραση. απόφαση δεν έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, είμαστε να τη λάβουμε υπόψη και θα είμαστε έτοιμοι. Αυτό δείχνει τη γελιότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει γίνει έκκληση από τα Ηνωμένα Έθνη. Το ΝΑΤΟ όμω και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε αγώνα δρόμου ποιο θα φτάσει πρώτο. Ωραία, λέει ο πρόεδρο και αυτή ήταν η τελευταία. Ε, ο τελευταίο τόνο στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Παπόφσκι. Σας είχαμε πει πόσο μας είχε ενοχλήσει η κατάσταση πριν από τρεις εβδομάδες. Εγώ προσωπικώς ε, ε το είχα εκφράσει ξεκάθαρα. Σήμερα είμαι κάπως ε, δύσθυμος. Μας είχατε μιλήσει πριν από τρεις εβδομάδες για μια προσεκτική για ένα προσεκτικό σχεδιασμό. Τώρα βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να ληφθούν πολιτικέ αποφάσει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην είμαστε έτοιμοι ω προ τον προγραμματισμό Εντάξει, η πολιτική απόφαση των κρατών μελών στη συνέχεια θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Θα είναι περίπλοκο να ληφθεί, θα πρέπει να είναι προσεκτική η εξέταση, θα υπάρξουν πολλέ αποκλίνουσε απόψει και όλα αυτά. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Αλλά εδώ και τρει εβδομάδε πώ είναι δυνατόν να μην γίνει το προγραμματισμό. Να μην έχετε προχωρήσει λίγο περισσότερο σε σχέση με αυτά τα οποία μα λέτε. Γι' αυτό που σα λέω, είμαι και απεσιόδοξο. Και ελπίζω όταν πια έχει τελειώσει αυτή η κρίση και έχει προχωρήσει ο προγραμματισμός και μάλιστα αποδειχθεί αποτελεσματικός. Ελπίζω να μπορούμε να τα πούμε διαφορετικά. Για τη εθνική απόφαση ήταν ουσιαστικά εκείνη η οποία έβαλε σε τέλος την κρίση. Και με τη μισράτα φαίνεται ότι το ίδιο θα γίνει τελικά. Θα χρειαστεί να παρισπίσει κάποια εθνική απόφαση για να τεθεί ένα τέλος στην κρίση. Όλες λοιπόν οι διαδικασίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ε, έχουν τελικά κάποιο νόημα, διαρωτώ με. Και όπως είπα, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ε, δυσκολίες ε, ως προς τη λήψη της πολιτικής απόφασης, αλλά, εν πάση περιπτώσει, προγραμματισμός θα μπορούσε ήδη να υπάρχει. Ευχαριστώ και εις το επανειδήν. Και τώρα η κυρία Αρνού παρακαλώ. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Είναι εδώ μαζί μας ε, η Claude France Αρνού, ε, η οποία μόλις ε, διορίστηκε εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Σας ομολογώ ότι θα ήθελα με την προηγούμενη της ιδιότητας ε, να την ε, ε, υποδεχόμαστε σήμερα. Επειδή ο προγραμματισμός μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ορισμένα πράγματα και με την προηγούμενη σας ιδιότητα. Όχι, λέει η κυρία Νου, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάπως απογοητευτήκαμε από τις ε, ε απαντήσεις που ακούσαμε από τον ε, ε κύριο Ποπόφσκι. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε και επίση ορισμένα πράγματα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, να μας πείτε και για τα προβλήματα προϋπολογισμού που αφορούν όλα τα κράτη-μέλη και που φυσικά είναι εμφανή σε όλα τα προγράμματα και σε όλες τις πολιτικές. Ε, ενδεχομένως να ε, μπορείτε να παίξετε έναν ε, διαφορετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτής της κρίσης που φαίνεται ότι θα διαρκέσει. Ίσως και εσείς ε, να μας πείτε περισσότερα για το ρόλο που πιστεύετε ότι θα διαγραμματίσει ο οργανισμός του οποίου είστε επικεφαλής. Ε, να μας πείτε και ορισμένα πράγματα για τον προϋπολογισμό δεδομένου ότι δεν αλλάζει και πολύ. Ε, τις, ε, διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες ε, με, για τη συνεργασία με άλλους ε, φορείς όπως για παράδειγμα το ΝΑΤΟ και κάποια προγράμματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί να μας πείτε ενδεχομένως ορισμένα πράγματα ε, μετά από την πρώτη εικόνα που έχετε πλέον διαμορφώσει στο πρώτο αυτό διάστημα της, του αξιώματός σας. Ευχαριστώ πολύ είναι ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη τιμή για μένα να είμαι και πάλι εδώ, βέβαια με διαφορετική ιδιότητα αυτή τη φορά. Φυσικά καλύτερα να μην σφετεριστώ εξουσίες που δεν έχω πια, Οπότε δεν θα σας πω τίποτα για το προηγούμενο μου αξίωμα. Θα προσπαθήσω λοιπόν όλη μου την ενέργεια να την συγκεντρώσω ε, για να υπηρετήσω τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Πρόκειται για ζητήματα βέβαια τα οποία είναι λιγότερο καυτά, λιγότερο δραματικά, λιγότερο άμεσα, αλλά φυσικά πρέπει το αύριο να προγραμματίζει κανείς και μάλιστα μερικές φορές ε, υποστηρίζοντας και ήδη δρομολογηθέντα προγράμματα και ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα όπως αυτά που ε, συζητάτε ε, σήμερα Νομίζω ότι φυσικά αυτό είναι και ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Όταν υπάρχει μια κρίση, έχει αντίκτυπο και στον προπολογισμό, είπατε και εσείς, το είπατε κι εσείς. Συνεπώς, το πλαίσιο που αναφέρατε κι εσείς, ε, δηλαδή τη μείωση του προπολογισμού. Ε, είμαστε πολύ κάτω από το 2% για πολλά κράτη-μέλη, ένα ποσοστό που είχε θεωρηθεί ε, ένας, ένα αρκετά καλό ποσοστό για την άμυνα σε εθνικό επίπεδο. Σε μια χρονική στιγμή, και αυτό το έδειξε και η σημερινή σας συζήτηση, που το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, οι απειλές, τα σενάρια αποσταθεροποίησης ε, δεν μειώνται. Και βέβαια σε μια χρονική στιγμή άλλα δραματικά σενάρια ε, διαφαίνονται, μπορεί να χρειαστούν και, στρατιωτικ... και στρατιωτικά ζητήματα αλλά και για προστασία των αμάχων, Λιβύη, Ιαπωνία, ε, βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί σε ένα, το τι μπορεί να συμβεί λόγω ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Ε, όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ανεξαρτήτως ε, της κρίσεως για την οποία συζητούμε κάθε φορά χρειαζόμαστε και στρατιωτική ε, ε, ικανότητες αλλά και άλλου είδους παρεμβάσεις, όχι απαραίτητο στρατιωτικές. Επομένως, μειώνονται οι αμυντικοί προϋπολογισμοί, ε, οι κρίσεις είναι όλο και περισσότερες, ε, παρεμβάσεις που δεν είναι υποχρεωτικά στρατιωτικές, το βλέπουμε και στη διαχείριση των κρίσεων, αλλά και στις διάφορες υποδομές. Ε, ενδιαφέρει λοιπόν αυτό ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις και όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε έχουν να κάνουν και με, το, και με, το, με την προστασία των αμάχων και με την τεχνολογία και με στρατιωτικά ζητήματα, με την ε, ε, εποπτεία ε, στις θάλασσες γιατί αναφερθήκατε και σε αυτό το θέμα ε, είναι όλα αυτά λοιπόν ε, τομεί ε, που είναι και στρατιωτικοί από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη πλευρά αφορούν ε, και τους πολίτες. Στο πλαίσιο λοιπόν που και εσείς αναφέρετε, ένας ανανεωμένος ρόλος για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ο οποίος είναι πολύ νέος, έξι ετών μόλις, διασώθηκε από τις συνθήκες, άρχισε να ισχύει πριν την έναρξη ισχύω τελευταία συνθήκης, εγώ ουσιαστικά αναλαμβάνω έναν οργανισμό ο οποίος ήδη υφίσταται και που έχει ήδη μία ομάδα, έχει πολλές ομάδες μάλιστα που λειτουργούν ε, και πρέπει να το πω αυτό γιατί η προκάτοχή μου το κατάφεραν αυτό, όχι εγώ, δουλεύει καλά η ομάδα. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ καλό μέσο, μικρό, είναι μικρό, ε, πολύ ε, συνεκτικό με έναν πολύ συγκεκριμένο προπολογισμό και ούτως ή άλλως θα σας πω και περισσότερα πράγματα όπως μου ζητήσατε για το θέμα του προπολογισμού. Όλα αυτά λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας, ε, να προσπαθήσουμε να έχουμε δομέ όσο το δυνατόν πιο ε, στεναρές αλλά όσο και πιο λιτές και νομίζω ότι ο οργανισμός μου πραγματικά τα καταφέρνει πολύ καλά. Από την άλλη, οι εταίροι μα στι Βρυξέλλε έχουν πολλά προβλήματα με αλλαγέ που πρέπει να γίνουν. Εμεί δεν έχουμε τέτοιου είδου πρόβλημα και δεν χρειάζεται να. Ε, είμαστε ακόμη πιο λιτοί από ό,τι ε, είμαστε τώρα. Και αυτό είναι πραγματικά ευτυχές. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Μας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουμε κατά παραγγελία, δηλαδή όταν χρειάζεται να είμαστε 26 ε, δουλεύουμε στα 20, με, 20, με 26 ε, μέλη, ε, όπως για παράδειγμα για πολύ σοβαρές έρευνες, για ζητήματα τυποποίησης, πιστοποίησης. Είναι καλύτερα να δουλεύουμε σε επίπεδο 26 κρατών μελών, γιατί είναι προστιθέμενη αξία όταν είμαστε περισσότεροι. Μερικές φορές όμως ξεχνάμε ότι ο οργανισμός δίνει τη δυνατότητα εργασίας ε, στον αριθμό των κρατών μελών που είναι έτοιμα να το κάνουν. Δύο, τρία, τέσσερα, όσα είναι, εν πάση περιπτώσει. Όμως, η δομή του οργανισμού, ε, για παράδειγμα τα προγράμματα κατηγορίας Β, έχουμε τη δυνατότητα μερικές φορές ε, να ε, αφορούν οι συζητήσεις τα προγράμματα των κρατών μελών που είναι έτοιμα να διαθέσουν τους πόρους και που έχουν ανάγκη τις συγκεκριμένες τεχνολογίες και θέλουν να διαθέσουν τους πόρους για να τις αναπτύξουν. Είμαστε λοιπόν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που προσπαθεί να λάβει υπόψη αυτή τη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας, δουλεύει κατά και παραγγελία και εξυπηρετεί τα κράτη-μέλη. Το είδα αυτό λοιπόν στη πρώτη εικόνα που διαμόρφωσα για τον οργανισμό. Τα, η, τα θέματα τα στρατιωτικά είναι καθαρά εθνικής κυριαρχίας, είναι κάτι το οποίο είναι αναμφισβήτητο. Εκεί είναι ο οργανισμός για να προτείνει, για να ε, συνεπικουρεί, αλλά σε καμία περίπτωση για να κάνει τον προγραμματισμό τον αμυντικό ε, αντικαθιστώντας τα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε πολλές φορές... Για παράδειγμα το dating agency λέγαμε συχνά δεν νομίζω ότι είναι και ο κομψότερος όρος θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει Εντάξει, τώρα αυτό εξαρτάται και από τα ε, είδη και έθιμα του καθενό, αλλά πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα χώρο που τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, συναντιούνται, να ε, συνεργάζονται για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Νομίζω λοιπόν ε, ότι αυτό που οθεί σε μια ανανέωση του ρόλου του οργανισμού είναι αυτό που είπατε ότι οι Υπουργοί Άμυνας το είπαν αυτό στη Γάνδη κατά τη Βελγική Προεδρία μείωση των πόρων τους και επομένως η προτεραιότητα λόγω της κατάστασης των, ε, της οικονομικής ε, αλλά και της διεθνούς συγκυρίας να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Οπότε αν με ρωτάτε ποιες είναι οι προθέσεις μου στο πλαίσιο αυτής της ε, κατάστασης είναι ότι η βασική προτεραιότητα είναι να βοηθήσει ο οργανισμός σε αυτή την προσπάθεια pooling and sharing. Ε, είναι λοιπόν αυτό πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς είναι κάτι που το κάνουμε πολλά χρόνια. Υπάρχουν ε, πολλά παραδείγματα. Κάθε φορά που θέλουμε να πούμε κάτι για τον οργανισμό, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για, για, για παράδειγμα, η επάνδρωση των ελικοπτέρων. Για, τα ελικόπτερα είναι ένα από τα βασικά ε, κενά των επιχειρήσεων είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στο ΝΑΤΟ. Όταν λοιπόν προτείνουμε και οργανώνουμε ασκήσεις μεταξύ των κρατών μελών για την ε, ε, εκπαίδευση των ελικοπτέρων σε ένα συγκεκριμένο ύψος ε, ή για την ταχύτητα ανάπτυξή τους, ε, για παράδειγμα στο Αφγανιστάν, κάνουμε pooling and sharing σε επίπεδο εκπαίδευσης. Το ίδιο κάνουμε και στο πλαίσιο της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολύ συγκεκριμένα και πολύ αποτελεσματικά. Δηλαδή, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού οργανισμού έχουμε δραστηριότητες ε, με κυρίαρχο τρόπο τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν πολύ συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες. Όλες αυτές λοιπόν οι ασκήσεις εκπαίδευσης προσπαθούμε να τις επεκτείνουμε και στα πληρώματα του Αφγανιστάν όπως κάναμε και με τα δικά μας πληρώματα ε, και αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της ε, συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ένα ακόμη παράδειγμα, pooling and sharing. Ε, όταν, ε, για παράδειγμα, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα εργαστήριο εγκληματολογικό, για την ε, τρομοκρατία, για παράδειγμα, επί τη βάση ενός συμβολέου που είχαμε ε, με μία ισπανική ε, εταιρεία η Ισπανία την ανέπτυξε αλλά η Γαλλία θα την αναπτύξει περαιτέρω. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε μια κοινή ανάλυση ε, μεταξύ Ευρωπαίων για να έχουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο εγκληματολογικό εργαστήριο και αυτό ε, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο μέτωπο του Αφγανιστάν αλλά και σε άλλα μέτωπα. Έχουμε και άλλα λιγότερο ελκυστικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν ε, καλύτερες ε, λύσεις ε, επιμελητίας. Προσπαθούμε να κάνουμε και πολύ σοβαρή αποταμίευση και σε θέματα επιμελητείας και στον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε άλλα προγράμματα συνεργασίας και έτσι να απελευθερώνουμε πόρους για περισσότερα προγράμματα. Δεύτερη προτεραιότητα που δεν είναι πάρα πολύ θεαματική αλλά είναι σημαντική γιατί οι Υπουργοί Άμυνα ε, προσπάθησαν να μας πούν τις προτεραιότητες τους ε, στο πλαίσιο ενός προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλιά το λέγαμε κοινοτικό πρόγραμμα αυτό, ένα λοιπόν που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό είναι του ενιαίου ουρανού με το πρόγραμμα Σεζάρ. Ένα πρόγραμμα που πραγματικά ε, θα αλλάξει εκ την ευρωπαϊκή αεροπορία, θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για τους Υπουργούς Άμυνας και από απόψεως ε, εξοπλισμού και από απόψεως διαδικασίας. Αυτό που περιμένουν ε, από εμά οι Υπουργοί και δεσμευτήκαμε να το κάνουμε και έχουμε κάνει και όλες τις απαραίτητες επαφές με τους συνομιλητές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ Θέλουμε λοιπόν όσο το δυνατόν περισσότερες συνιστώσεις ε, να τις λάβουμε υπόψη ε, και σκεφτόμαστε και τους χρήστες στα κράτη-μέλη που θα πρέπει όλα αυτά να τα μεταφράσουν σε εξοπλισμό στο μέλλον και να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στο πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ γιατί δεν είναι μόνο ένα ε, ζήτημα του τι θέλουν οι Υπουργοί Άμυνα, είναι και του τι επιπλέον μπορούμε να πετύχουμε στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού και στις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ Προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες του ΝΑΤΟ σε αεροπορικά ε, ζητήματα. Τα CD7 ε, για παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε, ή τα WACS, ε, προσπαθούμε να τα λάβουμε υπόψη. Να λάβουμε υπόψη και τους εθνικούς χρήστες, αλλά και να λαφθούν υπόψη οι ανησυχίες του ΝΑΤΟ στο στρατιωτικό επίπεδο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ο τρόπος ε, μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά δεν χρειάζεται να μπω σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ενδεχομένως ε, αν θέλετε να σας τις δώσω υπομορφή επιπρόσθετων πληροφοριών. Είναι σημαντικό πάντως να τις αναφέρω γιατί κάνουν, έχουν να κάνουν με πολιτικές για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα και την τεχνολογία. Είναι γεγονός ότι δεδομένη της κατάστασης μερικές φορές ε, ε, είμαστε λίγο επιπόλαιοι και υπάρχει περίπτωση, αν δεν κάνουμε τι απαραίτητε πρόοδου στην έρευνα και την τεχνολογία, να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα τελικά στους, ε, στους, στον αμυντικό μα εξοπλισμό. Και θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία, κυρίω για τι πιστώσει έρευνα ε, που είναι τμήμα του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου έχει νόημα, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασία. Υπάρχει άλλωστε ένα πλαίσιο συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σεβόμενο βέβαια τι επιλογέ που γίνονται από τη Δημοσιονομική Αρχή. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών προγραμμάτων και των στρατιωτικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, το διάστημα είναι ένα τομέα που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία που μόλι ανέφερα και στον τομέα τη έρευνα και τη τεχνολογία. Ένας ακόμη τομέας που αφορά και ε, άλλες ε, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ε, ραδι, οι, οι Και ένα τελευταίο στοιχείο για το οποίο θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με πλήρη σεβασμό των συνθήκων εφόσον η Ευρωπαϊκή, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, είναι ό,τι έχει να κάνει με την αγορά, το πακέτο της άμυνας και, και σε αυτό και για αυτό το θέμα η Υπουργοί Άμυνας επέμειναν στην καλή ερμηνεία και την καλή ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της ε, αγοράς και του ανταγωνισμού και από την άλλη των ιδιαιτεροτήτων και των χρήσεων ε, του άρθρου 346. Όλα αυτά πάντα σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επέμεινα πολύ σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και η πρότασή μου στην ύπατη ε, εκπρόσωπο, την κυρία Άστον, είναι νομίζω πολύ σημαντικό ε, να γνωρίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ε, οι Υπουργοί Άμυνας, ε, με τρόπο που να είναι αποτελεσματικό και για τους ίδιους. Θα ήθελα επίσης να αναπτύξω τις σχέσεις του οργανισμού με όλους τους σημαντικούς εταίρους του, στις διάφορες δομές του Συμβουλίου, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να συνεργαστούμε πολύ στενά. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνέχεια μεταξύ της ε, όλων των προσπαθειών στην ε, έρευνα και την τεχνολογία, όμως ε, εμείς ε, δεν είμαστε διαχειριστής των προγραμμάτων εξοπλισμών. Το, στη, στην καλύτερη περίπτωση να μπορούμε να πούμε την άποψή μας, όμως... Υπάρχουν και άλλα λοιπόν και άλλοι φορείς που είναι πολύ σημαντικοί για μας, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Διάστημα, της ε, ασφάλειας, ε, ε, της αεροπορικής ασφάλειας, με την οποία έχουμε ανανεώσει τις επαφές μας. Και κάτι ακόμη, ούτως ή άλλως σας είπα και πάρα πολλά παραδείγματα, που δείχνουν τη σημασία της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Υπήρχε ήδη μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ ημών και του ΝΑΤΟ ήδη όταν είχε ο προκάτοχός μου την εξουσία. Με τον στρατηγό Αμπριγιάλ ε, έχουμε συναντηθεί δύο, δύο φορές Είπα προηγουμένως για το ΣΕΖΑΡ, για τον ε, νιαίο ουρανό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνεργαστούμε με τους ε, ε γενικούς γραμματείς και τους αναπληρωτές γραμματείς. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συνεργασία μας ε, με το ΝΑΤΟ, μίλησα για την ε, σημασία των, ε, της καταπολέμησης χρήσης των εκρηκτικών μηχανισμών. Υπάρχουν τέτοιου είδους τομείς για τους οποίους θα χρειαστεί να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο με τον ΝΑΤΟ στο μέλλον, με σκοπό την προστασία των πολιτών. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και που φάνηκε από τις επισκέψεις που λάβαμε ήταν η σημασία των τρίτων εταίρων. Είδα πάρα πολλές επισκέψεις, είχαμε πολλές επισκέψεις από τη Ουάσιγκτον. Ε, το νούμερο 2 του Πενταγώνου ήρθε δύο μέρες μετά που διορίστηκα για να συζητήσουμε και είχε έρθει και στον οργανισμό για να δει ακριβώ ποιο είναι ο ρόλο του οργανισμού. Και από τότε έχουμε πολλέ επισκέψει από τη Ουάσιγκτον, τακτικέ για τα ζητήματα, για παράδειγμα, των εξαγωγών που ήρθαν ε, γνωρίζοντας βέβαια και τα συμφέροντά τους να δουν ε, πώς ακριβώς ε, δραστηριοποιείται ο οργανισμός, για παράδειγμα, σε ζητήματα εξαγωγών. Και η Ουκρανία και πολλοί άλλοι εταίροι εμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Θα προτιμούσα να σταματήσω εδώ αν συμφωνείτε, γιατί νομίζω ότι έχετε και ερωτήσεις, ενδεχομένως και κάποιες αμφιβολίες. Είναι η πρώτη φορά που ε, στην καριέρα μου νιώθω ότι το να επικοινωνεί κανείς είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ, δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι μας, ότι μας κατηγορούν ότι ε, υπάρχει κατακαιρματισμό των προσπαθειών. Είναι γεγονός όταν ερχόμαστε από μια χώρα όπω το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ζητήματα όπω αμυντικά προγράμματα ε, πρέπει να καλύπτουν τα πάντα. Οπότε ξεκίνησα και εγώ με αυτή την ε, ιδέα στο μυαλό μου και ενδεχομένω να τα λέω κάπω αδέξια, αλλά είναι γεγονό ότι πρέπει να τα καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θα κάνουμε προστασία του κυβερνοχώρου, α πούμε, αλλά θα ξεχάσουμε την προστασία του στρατιώτη. Δεν πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα παράλληλα, να είμαστε ορατοί και δεν είναι δυνατόν να ε, ε διασπαθίζονται και όλα οι πόροι. Έχουμε λοιπόν πολύ μικρό προπολογισμό, 30 εκατομμύρια ευρώ, 9 εκατομμύρια ευρώ επιχειρησιακού προποτορισμού. Θα ήταν καλύτερο να είναι μεγαλύτερο. Ε, αυτό πρέπει να πει ε, μια διευθύντρια ενό οργανισμού. Αυτό το έχω μάθει πλέον. Ίσως θα πρέπει να έχουμε περισσότερους σπόρους στη διάθεσή μας, ε, ειδικότερα για πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. Χρειαστήκαν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ 200 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, διατέθηκαν από τα κράτη-μέλη για, πολύ συγκεκριμένα για πολύ συγκεκριμένα προγράμματα και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί γιατί τα κράτη-μέλη σημαίνει ότι ε, διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το οποίο θα άξιζε τον κόπο να συγκεντρώσουν τους πόρους. Όταν λέω λοιπόν επικοινωνία, δεν είναι μόνο να λέει κανένας απλώς ε, πράγματα, σημαίνει αλληλεπίδραση μεταξύ ημών και των εταίρων μα, όλων των εταίρων μας. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ, όπως είπα και προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλέ επαφέ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εκπροσώπου όλων των κλάδων που μα ενδιαφέρουν και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί τη επιτυχία μα και θα θέλαμε πάρα πολύ να διατηρήσουμε αυτό το διάλογο μαζί σα. Ευχαριστώ. Euh, σα ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην Επιτροπή μας ε, να έχουμε συχνές επαφές έως των δυνατόν πιο συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων ε, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Πριν δώσω το λόγο στους αδέλφους, ε, Θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα και μην δυσαρεστείτε μαζί μου, δεν θέλω πολιτική απάντηση. Ξέρουμε για τη συμμετοχή στον οργανισμό πόσο σημαντικά πράγματα διακυβεύονται, ιδίω σε σχέση με την Τουρκία. Δεν θέλω, επαναλαμβάνω, να μου απαντήσετε συγκεκριμένα στο ερώτημα, αλλά σε σχέση με αυτή την τουρκική βοήθεια. Ποιε είναι οι τρίτε χώρε. Έτσι, μια, ε, έναν απολογισμό να μου κάνετε. Ποιε χώρε συμμετέχουν σε εργασίε του οργανισμού. Μιλήσατε για εταιρικέ σχέσει, είπατε για ενδιαφέρον τρίτων χωρών, αλλά συγκεκριμένα για μια τρίτη χώρα, όταν έχει καθεστώ παρατηρητή ή ε, συμμετέχει στον οργανισμό, τι κάνει ακριβώ, ε, για ποιε δραστηριότητε μιλάμε. Απάντηση. σα ευχαριστώ πολύ που πλαισιώσατε κατά αυτόν τον τρόπο την ερώτηση. Τρίτες χώρες οι οποίες συμμετέχουν ε, με διοικητική ρύθμιση, ουσιαστικά είναι μία, είναι η Νορβηγία η χώρα αυτή είδα πολύ συγκεκριμένα πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μόλις ανέλαβα το, τα καθήκοντά μου, έχουμε την Διευθύνουσα Επιτροπή, έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, 26 κράτη-μέλη που συμμετέχουν. 26 δηλαδή πλήν της Δανίας. Και έχουμε και μια ειδική συνεδρίαση με την Ορβηγία μαζί. Και έχουμε και τη δυνατότητα υπό την επιφύλαξη να γίνει αποδεκτό αυτό από τα κράτη-μέλη, να καλέσουμε την Νορβηγία και σε κάποιες από τις συζητήσεις μας. Η Νορβηγία λοιπόν, όπως και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Πατρίκ Ορουά, και η Νορβηγία είχαν προσκληθεί σε κάποιες συναντήσεις μας για ένα-δυο συγκεκριμένα θέματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη φάση που ελπίζω σύντομα να ολοκληρώσουμε μια αντίστοιχη συμφωνία με την Ελβετία, στο πέρα μια πάρα πολύ ε, μακρά και δύσκολη διαδικασία, ενώ δεν υπήρξαν πολιτικά ε, κολλήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πολύπλοκε διαπραγματεύσει ούτω ή άλλω. Εσεί αναφέρατε την Τουρκία Ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσει στον οργανισμό έχουν ολοκληρωθεί και το θέμα τώρα είναι στο Συμβούλιο, άρα για μένα εντάξει δεν είναι πρόβλημα να μιλήσω, ε, είμαι σε αρκετά ε, εύκολη θέση, αλλά έχω συναντήσει και εγώ τον πρέσβητη τον Τούρκο και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κάποιες επαφές. Ε, το ίδιο έκανα και στην προηγούμενη μου θέση, στην Διεύθυνση για τη Διαχείριση Κρίσεων και για το Σχεδιασμό. Το ίδιο πρέπει να σας πω ότι είναι σημαντικό ε, συνομιλητής μας Τουρκία ό,τι αφορά τις δυνατότητες. Όταν έχουμε ρεαλισμό και καλές προθέσεις μπορούμε να συνεργαστούμε. Και άλλα κράτη έχουν, ε, δείξει, ε, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Ουκρανία, επί παραδείγματι. Και χθε, εντάξει, όχι χθε, πολύ πρόσφατα, ο Σέρβος Υπουργό Άμυνα εξέδηλωσε και αυτό ενδιαφέρον. Αυτά προ το παρόν. Αυτό είναι ο κατάλογο. Έχουμε βέβαια συμφωνίε και με τρίτε οργανώσει, ΚΑΡ, ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό διαστήματο. Πολύ σύντομα ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει και με αυτού τους φορεί τη συμφωνία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις αυτές. Η Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ για τα όσα μας λέτε. Χαίρομαι που σας βλέπω κεφαλής της υπηρεσίας. Πρέπει να σημειώσω ότι έχω εξαίρετη εμπειρία συνεργασίας με την υπηρεσία. Όταν χρειάστηκε να σας συναντήσω για μια έκθεση ε, για το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών ε, ε, πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών καταστροφών. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχετε τουλάχιστον αυτό το επικοινωνιακό ταλέντο που χρειάζεται, όπως είπατε, η υπηρεσία. Θα υπενθυμίσω επίσης ότι όταν ήρθε για το, η ακροασή η κυρία Άστον, προκειμένου να εξασφαλίσει την επικύρωση της στη θέση του ε, εκπροσώπου, της έδωσα μια ερώτηση για την υπηρεσία της, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και τη ρώτησα συγκεκριμένα εάν μπορούσε να δεσμευθεί ως Βρετανίδα ότι θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί σε επίπεδο υπηρεσία, πολίτη, προπολογισμού και όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορέσει η υπηρεσία να αυθυγραμμιστεί στην εργασία των λοιπόν θεσμικών, των θεσμικών οργάνων και κυρίως των υπουργών ε, αμήνες. Η κυρία Άστον φαίνεται όμως ότι στα αγγλικά δεν μπόρεσε να πιστεί για αυτό το σκοπό. Ερωτώ λοιπόν τώρα, επ' αυτή σας την ιδιότητα, τώρα που είστε κεφαλής αυτής της υπηρεσίας, βλέπετε κάτι να έχει αλλάξει. Συμφωνία που πρόσφατα υπέγραψαν ε, η Γαλλία με την ε, Μεγάλη Βρετανία, κυρίως με την ιδέα του pooling και sharing πόρων ήδη βλέπετε να έχει εφαρμογή και σε επίπεδο υπηρεσίας. Δηλαδή υπάρχουν αιτήματα προς την υπηρεσία για νέες ιδέες, για σχέδια συγκεκριμένα που θα εξορθολογήσουν ενδεχομένως κόστος και έτσι θα επιτρέψουν την ε, μετατροπή των κονδυλίων αυτών σε κονδύλια που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για, τα, για τις πραγματικές μας ανάγκες. Αυτά που ονομάσατε και εσείς νωρίτερα, περιπτώσεις που δεν είναι μόνο στρατιωτικές ανάγκες, αλλά και μη στρατιωτικές πολιτικές. Ευχαριστώ κύριος Μπιτσικόφερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στον όλο αυτό το τομέα της πρωτοβουλίας από τη Γερμανία και τη Σουηδία για το pooling και sharing στο πλαίσιο της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, ασφάλειας και άμυνα, συγγνώμη. Και να ρωτήσω εάν βλέπετε πως έχει προχωρήσει η αποτελεσματικότητα χάρη στη συνεργασία ή όχι. Διαβάζω ότι η EDA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, σε μια σε ένα ανακοινωθέν τύπου είχε αποδώσει σε αυτή την πρωτοβουλία πολύ μεγάλη σημασία. Όμως δεν βλέπω από αυτά που λέτε εσείς να έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, να έχει πέσει μεγάλο ρόλο στις εργασίες της. Είπατε, μάλλον δόθηκε η εντύπωση από αυτά που είπατε, ότι μπορεί να κατακαιρματίζεται η υπηρεσία. Ε, εν πάση ελπίζω να μην είναι σωστό αυτό, αλλά υπάρχει κάτι που αντιμετωπίζει την, τον ενδεχόμενο κατακαιρματισμό. Και τα κράτη-μέλη έχουν πράγματι την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να συνεργαστούν στο πλαίσιο αυτής της Βλέπουμε τη συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, σε παραδείγμα, την αναπτύσσεται εκτός της υπηρεσίας και σε διαφορετική κατεύθυνση. Προφανώς υπάρχουν και πολιτικές ε, αντιρρήσεις ή ζητήματα που θα πρέπει κανείς να επεξεργαστεί. Θα ήταν καλό να μας τα εξηγήσετε πιο περιγραφικά και κυρίως αυτό που είπατε σε μια ε, συνέντευξη τύπου ότι αποτελεί προτεραιότητα αλλά δεν το παρουσιάσατε εδώ τουλάχιστον. Και επίσης συμπληρώνω ότι αναπτύξατε τις θέσεις σε μια σειρά θεμάτων μέχρι και τις ραδιοσυχνότητες, μέχρι και θέματα πολιτικής βιομηχανίας, θέματα για τα οποία εγώ δεν αναγνωρίζω προτεραιότητες, τουλάχιστον στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας σας. Μπορείτε να με διαφωτίσετε λίγο περισσότερο. Και τελευταία παρατήρηση. Έρευνα. Μιλήσατε για την έρευνα και το πόσο καταπληκτικό πράγμα είναι η υπηρεσία για την άμυνα να μπορεί να αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ε, αποφασίστηκε όμως αυτήν την εβδομάδα ότι δεν είναι μεταξύ των καθηκόντων της υπηρεσίας σας και προφανώς είστε ήδη ενήμεροι. Αν όμως έρχεστε να μας παρουσιάσετε ένα τέτοιο σχέδιο ή εγχείρημα το οποίο τόσο πολύ σας ενδιαφέρει, πώς μπορείτε να πείσετε το Κοινοβούλιο και την Ολομέλεια. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ε, τη δυσφορία της υπηρεσίας σας, διότι τα κράτη-μέλη ε, προφανώς δεν ε, προάγουν αρκετά αυτό το καθήκον, το οποίο ως αρμοδιότητα θα ανήκε στα ίδια, ενώ εσείς από την άλλη πλευρά έχετε λάβει υποστήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν καταλαβαίνω γιατί αντί να επιμείνετε και να πιέσετε για αυτό το οποίο ακριβώς σας ενδιαφέρει και το οποίο σε τελευταία ανάλυση ήταν και η δουλειά σας, ε, διαχέεστε σε άλλα πράγματα και δεν δίνετε έμφαση σε αυτό. Επίσης για την έρευνα ως προτεραιότητα θα πω ότι δεν έχω πιστεί διότι ούτε χρήματα έχουμε ούτε αρκετά μπορούμε να προχωρήσουμε στην συνεργασία σε επίπεδο υπηρεσία αμήνη μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή δεν βλέπουμε τα κράτη-μέλη νητεθειμένα να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν θα έλεγα να μην προσπαθούμε να χτυπήσουμε λάθο πόρτα, να επιμείνουμε, να επιμείνετε σε εκείνα τα θέματα που είναι δική σα αρμοδιότητα που μπορούμε από κοινού κατά τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό να υλοποιήσουμε. κυρία Αγνού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γκόμας. Είχα χτάνει την ευκαιρία να συζητήσω με την κυρία Άστον για την ε, κατάσταση, την κατεπίγουσα. Έχω την εντύπωση ότι μέσα σε αυτήν την πληθώρα συνεδριάσεων υπουργών στη Γάνδη και κυρίως στη Βουδαπέστη όπου συζητήσαν από κοινού τη μεγάλη ανάγκη για συνεργασία και κυρίως στην επίπεδο υπηρεσίας ε, αμήνης, δηλαδή να είναι σε θέση η υπηρεσία να επιτελέσει το έργο της για τις ε, δημοσιονομικές πτυχές. Πιστεύω ότι αν είχε σημαντικότερο προπολογισμό θα κάνει και πιο καλά τη δουλειά τη η υπηρεσία. Και μάλιστα και με πιο μακροπρόθεσμο όραμα, δηλαδή με ένα τριετή προπολογισμό. Βέβαια η κατάσταση οικονομική είναι αυτή που γνωρίζουμε όλοι μα. Και δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό, θα επεξεργαστεί βέβαια τι μεσονομικέ προοπτικές του Κοινοβουλίου Γέννη. Δεν ξέρω αν είναι πιο ρεαλιστικό να επιδιώξει κανεί τριετή προοπτικέ που σημαίνουν και πιο πολλά χρήματα. Πριν αποδεθεί κανεί σε μια μάχη, δηλαδή, καλό θα είναι να ξέρει που θα τον ευγάλει αυτή η μάχη, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση των πρωτομελών, Θα ήταν καλό να ξέρουμε αν θα είναι θετικό το αποτέλεσμα τη μάχη ή όχι. και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς με τις δυνατότητες που έχουμε στο πλαίσιο του pooling and sharing και στο πλαίσιο της υπηρεσίας. Ε, επίσης μιλήσατε για την ε, γάλλο-αγγλική συνθήκη. Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο την υπηρεσία. Είναι θέμα ιστορικής πολιτικής, αλλά θα επισημάνω ότι μόλις, μόλις διορίστηκα με καλέσε η Βρετανία πρώτη να συζητήσουμε για να κάνουμε κάτι το ρεαλιστικό και το αποτελεσματικό. Αλλά όπως είπα, ιστορική πολιτική είναι αυτή που είναι και εγώ δεν είχα λόγο να μιλήσω. Απλώς ό,τι μπορούμε από πλευρά μας για αποτελεσματική δουλειά, για δουλειά που ανταποκρίνεται στις ανάγκες, το πράττουμε. Ήγαλο, αγγλικη τώρα συνθήκη. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Φερρυπίν ο των ρηχείων, όπως λέμε. Υπάρχει κάτι το οποίο η Γαλλία με τη Βρετανία αποφασίζουν να πράξουν από τις από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για το θεωρούν σημαντικό και με συγκεκριμένη περιγραφή γιατί ανταποκρίνεται σε κάποιες συγκεκριμένε ανάγκες στις οποίες έχουν, δώσει απόλυτη έχουν αποδώσει απόλυτη προτεραιότητα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο να επιτρέπει και στα άλλα κράτη-μέλη να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Πολλά λοιπόν είναι έκρημη και όχι μόνο στο επίπεδο και, και Γάλλων. Και εμείς από την υπηρεσία πρέπει να πιέσουμε δε και άλλα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στα σχέδια αυτά τα εγχειρήματα και τη τεχνολογία. Το ότι πρόκειται για Γάλλο-Βρετανική συνθήκη δεν με αφήνει παρά να κάνω τα εξή σχόλια, ότι υπήρξε μια άνωθεν πολιτική βούληση, ένα, και η δέσμευση ότι θα υλοποιηθεί αυτό με τη χρηματοδότηση κτλ. Το ίδιο λοιπόν θα μπορούσε να κάνει και η υπηρεσία μα, εάν υπήρχε η πολιτική βούληση και η δέσμευση που θα μα διαθέτει και τα κονδύλια. Ε, το ίδιο και για σχέδια που μερικέ φορέ έχουν ή για έργα, τα οποία μερικέ φορέ έχουν και ζωτική σημασία αρκεί να υπάρξει ένα κοινόχρονο διάγραμμα. Και όταν η κατάσταση οικονομική είναι πιο κατάλληλη, ίσως αυτό δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσει και τον κύριο Πιτικόφερ, ε, εάν λοιπόν είναι πιο κατάλληλη η χρονική στιγμή και επιτρέπει περισσότερη συνεργασία. Αν είναι τώρα κατάλληλη, πάντως τα κράτη δεν το, δεν το μετατρέπουν σε πράξη αυτό που καμιά φορά λένε ότι δηλαδή είναι η συγκυρία ε, κατάλληλη. Ε, στα γερμανικά ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω γερμανικά όπως ο συνάδελφος νωρίτερα δεν θα τα καταφέρω. Συνεχίζω στα γαλλικά. Η υπηρεσία έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για το polling and sharing. Η γερμανο-σουηδική πρωτοβουλία είναι μια πρόσθετη πολιτική πρωτοβουλία, πολύ σημαντική δεν την κατέγραψα εγώ ως πρωτοβουλ... πρωτο... προτεραιότητα, γιατί και βέβαια πρέπει η υπηρεσία να συμβάλλει, αλλά υπάρχει και πολλή δουλειά στο πλαίσιο της ε, στρατιωτικής επιτροπής και σε αυτό επέμειναν ιδιαίτερα οι Γερμανοί και οι Σουηδοί, δηλαδή να επεξεργαστεί το θέμα η στρατιωτική αυτή επιτροπή και να δουν τι μπορούν ως pooling και sharing να προσφέρουν τα κράτη. Και αυτό θα έρθει στην επόμενη συνεδρία των Τσότ, των αρχηγών ε, επιτελείων, θα συζητηθεί αυτό και η βάση των ε, συμβολών ε, των κρατών μελών ε, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας Γερμανίας και της Σουηδίας τι μπορούν να προσφέρουν τα κράτη-μέλη. Πόρους και χρονοδιάγραμμα, στους οποίους δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Πολύ δουλειά λοιπόν υπάρχει ακόμη και ίσως να μην το εξεφράσα καλά νωρίτερα, ήταν η πρώτη προτεραιότητά μου το pooling and sharing. Αυτό ανακοίνωσα ω πρώτη προτεραιότητα. Και αν μπορούμε να δώσουμε και πρόσθετα μέσα για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό, πολύ ευχαρίστω. Δεν θα σας εκθέσω διάφορα σχέδια, αλλά στη Γαλλία τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχουν 3, 4, 5 έργα τα οποία έχουν προτεραιότητα. Και άλλωστε αυτό θέλουν και τα κράτη-μέλη. Θέλουν πρώτα να δουν κάποιο αντίκτυπο στο πλαίσιο το στρατιωτικό των συμβολών τους και στη συνέχεια ε, να ληφθεί η απόφαση για το τι, ποια σχέδια, ποια έργα θα στηριχθούν. Ένας υπουργό, Γάλλος τυχαίο. Ε, εξέφρασε με πολύ επιτυχημένο τρόπο ε, την κατάσταση στη Βουδαπέστη Είπε λοιπόν ότι δώσαμε για την υπηρεσία, ορίσαμε το μενού. Τώρα ήρθε η ώρα κάποιο να σερβίρει τα πιάτα και κάποιο να πληρώσει και το λογαριασμό. Είμαστε έτοιμοι ως προς την, την κουζίνα, την έχουμε έτοιμη, την έχουμε καθαρίσει, ετοιμάσει, έχουμε τα πιάτα έτοιμα για σερβίρισμα. Τώρα πια πρέπει να ληφθεί το επόμενο βήμα. Επίσης ξέρω και για τη συζήτηση στην ε, Επιτροπή ε, Ήτρε για την έρευνα. Δεν θα ήθελα τώρα να ε, συμμετάσχω στην συζήτηση που ανοίξει το κοινοβούλιο. Δεν πρέπει εγώ να κάνω τέτοια παρέμβαση. Για το υλικό διτής χρήσης, όταν μιλάμε για το διάστημα, δεν είναι ούτε στρατιωτικό ούτε μη στρατιωτικό. Όταν μιλούμε για θαλάσσια υποπτία ή επιτήρηση, ε, πολλές φορές είναι διπλής χρήσης. Όταν μιλάμε για drones, για μη επανδρομένα αεροπλάνα και γι' αυτό αναφέρθηκα και στον αντιδραστήρα τον Ιαπωνικό. Ο κύριος χρήστης του ανεπάνδρωτου αεροπλάνου μάλλον είναι το μη, το μη στρατιωτικό σκέλος. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε πολύ υλικό για το οποίο δεν είναι σαφές ότι είναι στρατιωτική χρήση ή μόνο στρατιωτική χρήση. Άρα δεν καταλαβαίνω αυτές τις επιφυλάξεις για το υλικό αυτό. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το σύνολο των χρήσεων που θα επιτρέψει αυτή η τεχνολογία στα κράτη-μέλη να συγκεκριμενοποιήσουν στη συνέχεια. Εγώ αυτό δεν ήθελα να το παρουσιάσω σαν ερζάς, σαν υποκατάσταση. Στην πραγματικότητα έχουμε περισσότερο να κάνουμε με pooling και sharing. Αλλά πάλι, όπως είπα, δεν αποφασίζω εγώ. Τα κράτη-μέλη θα ορίσουν το pool and share, θα διαθέσουν τους σπόρους και θα κάνουν αυτή την, ε, θα λάβουν αυτή την απόφαση όπως έγινε με την καλογερμανική συνθήκη άνωθεν και εμείς είμαστε απλώς έτοιμοι στην αφετηρία στις θέσεις μας όπως λέμε στον αθλητισμό για να ξεκινήσουμε τον αγώνα δρόμου. Ό,τι αποφασίζουν τα κράτη-μέλη όμως. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας για να τα στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Πάσκου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι και εγώ εξ αυτών που θέλω να σας καλωσορίσουν εδώ, κύριε Αρνού, και να σας πω ότι κάθε φορά που συναντώμαστε η συζήτηση που έχουμε είναι πάρα πολύ καλή και ενημερωτική, διαφωτιστική. Έχω ένα ενοιολογικό ζήτημα, έτσι θα το χαρακτήριζα. Στις αρχές του 2000 ξέραμε ότι με το Ιράκ διχάστηκε το ΝΑΤΟ και οι διατλαντικές σχέσεις. Μία, ένα από τα βασικά στοιχεία Ε, διχασμού αν θέλετε ήταν ακριβώς η ιδέα αυτής της, ε, του συνασπισμού της συμμαχίας των προθήμων. Και αυτή ακριβώς η έννοια ε, ήταν χώρες, οι πρόθυμες χώρες δηλαδή, οι χώρες που ήταν διατεθειμένες να συμμετέχουν σε μία περισσότερες δράσεις, κάποιες άλλες χώρες δεν ήταν διατεθειμένες. Η εντύπωση που έχω αποκομίσει εγώ είναι ότι τελικά Ακόμη και αν δεν μιλάμε ακριβώ για το ίδιο πράγμα, δεν είναι η ίδια έννοια ακριβώ, αλλά αυτό που κάνουμε το ίδιο είναι. Περί συμμαχία των προθύμων πρόκειται. Και συμμετέχουν οι χώρε που θέλουν να έχουν αυτή την ε, μόνιμη διαφορετική συνεργασία. Έχουμε συμμαχία των προθύμων, συμμαχία των προθύμων στη, στο ΝΑΤΟ τώρα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Αλλά και τώρα και στον οργανισμό έχουμε χώρες που δεν είναι πρόθυμες να συνεργαστούν για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λίγο πολύ δηλαδή έχουμε διάφορες μορφές συμμαχιών προθύμων. Είτε για κάποιες δράσεις, είτε για κάποια σχέδια, προγράμματα ή δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Είναι λοιπόν αυτός ένας τρόπος να μην υπάρξει εμπόδιο σε, στην ανάληψη κάποιων δράσεων. Αυτός, αν κάποιες χώρες θέλουν να λάβουν δράση να μπορούν. Και επόμενο ερώτημα, πώς αυτό θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της Ένωσης αυτής καθεαυτή όταν αρχίζουμε να επιτρέπουμε σε κάποιες χώρες να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτό το πλαίσιο των συμμαχιών ή συνασπισμών των προθήμων. Ας ε, πάρουμε ένα παράδειγμα. Κάποιες χώρες, σημαντικές, μεγάλες χώρες, σε συμμαχίες των προθήμων συμμετέχουν σε κάποιες δράσεις. Και έφνησε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση που ε, για αυτήν υπάρχει επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης. Και λέει μια χώρα, α, με συγχωρείτε, έχω αναλάβει ήδη πάρα πολλές υποχρεώσεις εκεί, εκεί και παραπέρα. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Άρα πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία. Πρέπει να εξορροπήσουμε αυτή την τάση που ε, υπαγορεύεται από την, ε, το ρεαλισμό. Κάποιες χώρες να θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη δυνατότητα ε, σεβασμού των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει χώρε στο πλαίσιο τη συνθήκη Αν αυτό τεθεί κάποια στιγμή. Αυτό ήταν το ενιολογικό μου, το ιδεολογικό μου ερώτημα. Απάντηση. Ωραίο ερώτημα πάντως. Αλλά δεν μπορώ να προσπιθώ ότι έχω και την απάντηση στο ερώτημά σας. Πρέπει να το σκεφτώ. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σας. Ε, πρώτη αντίδραση αλλά μάλλον θέλω να το σκεφτώ ακόμη περισσότερο. Ε, τέλος πάντων, η πρώτη μου αντίδραση είναι η εξή. Κάπως έτσι έχει λειτουργήσει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που είναι εντελώ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οργανισμός και με τις περιορισμένες μου αρμοδιότητες εκεί θα επικεντρωθώ. Αυτό που προσφέρει είναι η δυνατότητα επίτευξης συμβιβασμού, δηλαδή να έχουμε την οροφή ένα σημείο όπου εντός ενός θεσμικού πλαισίου, του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού στην περίπτωσή μας, του Συμβουλίου, αν θέλετε, να μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Άλλοτε, ε, κατά παραγγελία, άλλοτε από όλα τα κράτη-μέλη, τα 26 που είναι στον οργανισμό. Ίσως, ε, παραδείγματο χάρη, όταν μιλάω αλακάρτ. Κάποια κράτη-μέλη να μην θέλουν να δεσμευθούν όταν δεν είναι κοντά γεωγραφικά ε, το θέατρο επιχείρησεων κτλ. Για το Ιράκ, εντάξει, ήταν κάπως διαφορετικό. Ε, πάντως παίζει ρόλο η γεωγραφία, η ιστορία κτλ. Και πρέπει να βρούμε λοιπόν ε, κάποιο συμβιβασμό μεταξύ του κοινοτικού και του διακυβερνητικού επίπεδου. Υπάρχει αυτή η θεσμική οροφή κάτω από την οποία γίνονται κάποια πράγματα στον οργανισμό, αλλά είπα, σε κάποιες περιπτώσεις ε, και 26 χώρες, σε κάποιες άλλες 2-3 χώρες αλλά έχουμε αυτό το στοιχείο που δίνει ένα είδος συνεκτικότητα στον οργανισμό και τη δυνατότητα ε, της ε, συνεργασίας, ε, της ομαδοποίησης, να μην υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα του κατακαιρματισμού, της διασκόρπισης, της διασποράς των προσπαθειών και αυτό το θεσμικό πλαίσιο, αυτή, αυτός ο χώρος ο θεσμικός εξασφαλίζει και αυτή την εξισορρόπηση είπαμε, κάποια ε, αναλαμβάνουν κάποια μιλμόνο, σε κάποια άλλα θέματα καλό είναι να διατηρηθεί η συνέπεια, συνεκτικότητα και η αλληλεγγύα να γίνουν όλα σε επίπεδο των 26 χωρών μελών. Ο Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Διευθύντρια για την παρουσίαση, την πρώτη αυτή παρουσίαση. Θα έχουμε, ελπίζω, τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την εξέλιξη των διαφόρων προγραμμάτων, των συζητήσεων, των διαφόρων εταιρικών σχέσεων, των θεμάτων που άπτονται βέβαια και του προπολογισμού. Πάντοτε είστε ευπρόσδεκτοι στην υποεπιτροπή μα και ελπίζω να έχουμε πολλέ φορέ τη δυνατότητα να σα έχουμε εδώ για έναν επικοδομητικό διάλογο. Σα ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Bien, euh, nous poursuivons avec... Συνεχίζουμε με τον δεύτερο προσκεκλημένο μας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Μιώτσο, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Αντιμετώπισης Κρίσεων και Επιχειρησιακού Συντονισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα στην Υποεπιτροπή μας. Είναι η πρώτη σας παρουσία στην ε, Υποεπιτροπή μας. Ε, και θα θέλαμε να ακούσουμε ε, τη θέση σας, επειδή διαβάσαμε το οργανόγραμμα μεν της, ε, εξωτερικής, της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά θέλουμε να ξέρουμε περισσότερο για τον επιχειρησιακό χαρακτήρα των, της ιδιότητάς σας, να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τη Λιβύη, Είχατε πάει όλα στη Λιβύη, ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ. Είχαμε και μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ποπόφσκι στην αρχή της ε, σημερινής μας συνεδρίασης που μας ε, άφησε με πολύ περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Ελπίζω λοιπόν να έχετε κάποιες απαντήσεις να μας δώσετε. Το ελπίζουμε. Είναι ένα κατεπήγον ζήτημα και θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μας διαφωτίσετε. Θα θέλαμε μία πιο συνεκτική ε, συζήτηση για τη Λιβύη με ένα ενιαίο πάνελ, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι τα πράγματα τώρα. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα με ε, ίση σημασία όμως. Μήπως θα μπορέσετε κι εσείς, μήπως μπορείτε κι εσείς να μας πείτε ορισμένα πράγματα περισσότερα, πώς Διαχειρίζει το θέμα αυτό της Λιβύης ε, με την δική σας ιδιότητα. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντονζό. Θα σας μιλήσω για την επίσκεψή μου την περασμένη εβδομάδα στη Λιβύη και μέσα από την παρουσίασή μου αυτή θα σας απαντήσω ε, και σε όλα αυτά που με ρωτήσατε για το τμήμα το οποίο διευθύνω εγώ στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Την προηγούμενη εβδομάδα κατόπιν ετήματος της ΥΠΑ της εκπροσώπου στη Βενγκάζη. Για τρίτη φορά επισκέφθηκα τη Λιβύη. Μέσα στον ε, τελευταίο μήνα. Πρώτα πήγα στην Τρίπολη πριν από ένα μήνα, μετά στη Βενγκάζη, πριν από τρει εβδομάδε και δεύτερη επίσκεψή μου την προηγούμενη εβδομάδα στη Βενγκάζη. Η τελευταία τώρα αποστολή που είχα ήταν μια διυπηρεσιακή αποστολή ουσιαστικά. Ήμουν με μια δεκαμελή ομάδα ε, από την ΕΙΕ, την ΤΕΠΚΟ, την FBIS και την αντιπροσωπεία της Τινησίας και του Καΐρου. Πάρα πολύ σημαντικές ε, διπηρεσιακές συναντήσεις είχαμε με στόχο να κάνουμε μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης σε αυτό το τμήμα της Λιβύης και να προσδιορίσουμε δεχόμενες δράσεις που θα μπορούσε να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή. Στη Βεγγάζη συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Μουσταφά Λαμπτζεζαλίλ, τον πρόεδρο του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου, καθώς και με μέλη του Μεταβατικού Συμβουλίου, κάποια ως ακαδημαϊκούς, μέλη της πολιτών, με γυναίκες, με φοιτητές, με νέους, είχαμε επαφές και επίσης και, επίσης και με διπλωμάτες. Διπλωμάτες από τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τέσσερα κράτη-μέλη που έχουν παρουσία στη Βενγκαζιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Πολωνός ε, ε, πρέσβης στη Λιβύη, ο οποίος ε, είχε φύγει από την Τρίπολη και ήταν μαζί μας σε αυτήν την αντιπροσωπεία. Πριν πάμε στην Λιβύη, είχαμε συναντηθεί και με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών που ήταν στο Κάιρο, τον κύριο Καλίκοφ, συντονιστή ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Λιβύη. Και είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Κάλικοφ και κάποιους εξωματούχους από το Γραφείο των Προσφύγων και κάποιες άλλες υπηρεσίες των ΗΕ που εργάζονται ε, για ανθρωπιστικά θέματα σε σχέση με την κρίση στη Λιβύη. Στη Βεγγάζη συναντηθήκαμε επίσης και με τον απεσταλμένο τον ΙΠΑ, ε, τον κύριο Πρέντης. Κάποιες παρατηρήσεις για την ίδια την επιχείρηση, για την αποστολή ή τουλάχιστον τι εμείς ε, ε, τι εντύπωση αποκομίσαμε, πώς αντιληφθήκαμε τα πράγματα. Η κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη ξεκολουθεί να είναι απρόβλεπτη και ιδιαίτερα ρευστή. Με αυτά θέλω να σας πω ότι στη Φεγγάζη πραγματικά είχαμε την εντύπωση ότι εντός ωρών μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει μείζον ανθρωπιστική κρίση στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης. Οι εχθροπραξίες, οι στρατιωτικές είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένες, δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το επίκεντρο των συγκρούσεων. Η Μισράτα είναι μια πολιορκούμενη από τα στρατεύματα του Καντάφη πόλη και στο συγκεκριμένο μέρος αυτό, σε αυτή την πόλη, στο δυτικό μέρος της Λιβύης, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από ό,τι στο ανατολικό. Ξέρουμε ότι στη Μισράτα η καταστολή είναι πάρα πολύ έντονη. Έχουμε ελεύθερους έχουμε βομβαρδισμούς. Και χθες είχαμε κάποιες αναφορές ε, από την ICACP και το γαλλικό ε, Ερθρό Σταυρό που επισκέφθηκαν την πόλη στο κομμάτι που είναι κοντά στο λιμάνι. Μας είπαν πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά ε, μάλλον από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι σχετικά ηρεμή θα έλεγα, μάλλον δεν είναι αυτή η σωστή λέξη, γιατί υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές όπως σας είπα, υπάρχουν στρατεύματα τα οποία βρίσκονται 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η Ανατολική Λιβύη, όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, ε, βρίσκεται σε μία περίοδο έντονης δημοκρατικής επανάστασης. Φαίνεται ότι υπάρχει γνήσια επανάσταση, την οποία στηρίζει ο πληθυσμός ε, ευρύτατα. Τον στηρίζουν, τη στηρίζουν οι γυναίκες, οι νέοι, οι φοιτητές, οι διανοούμενοι και γενικά τα άτομα που εμείς συναντήσαμε στη διάρκεια της επίσκεψής μας εκεί. Θέλω να πω και να επαναλάβω ότι είχαμε την εντύπωση ότι ήταν ένα γνήσιο κίνημα επαναστατικό. Αυτή την εντύπωση αποκομίσαμε όλα τα μέλη της αποστολής μετά τις συναντήσεις που είχαμε με όλους όσους καταφέραμε να συναντηθούμε στη διάρκεια της αποστολής μας. Υπάρχουν στοιχεία ότι αναδύεται, εμφανίζεται μία κοινωνία των πολιτών που έχει κίνητρα ε, να αλλάξει τα πράγματα, έχει αποφασιστικότητα, αλλά δεν έχει εσωτερικό συντονισμό. Και ουσιαστικά δεν έχουν εμπειρία ε, διοικητική, εμπειρία διαχείρισης της κατάστασης. Αυτή η αναδυόμενη, όπως είπα, κοινωνία ε, των πολιτών, αναδυόμενη γιατί, σας είπα, μιλήσαμε με γυναίκες, μιλήσαμε με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, που πρόσφατα δημιουργήθηκαν και μας είπαν ότι επί δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν καμία ανθρωπιστική δραστηριότητα. Ούτε καν να πούν ότι μπορούν, βοηθούν κάποιον. Γιατί επί Καντάφη κανείς υποτίθεται ότι δεν χρειαζόταν ε, να λάβει κάποια υποστήριξη από την κοινωνία των πολιτών. Επομένω, αυξάνονται οι οργανώσει αυτές, ε, έτσι είναι αυθόρμητη η δημιουργία τους ε, και ο ρόλος ε, των γυναικών εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό το εκτιμά και το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο. Meeting with the, ε, ε, Mustafa Με τον Αμπτέλ Ζαλίλ, όπως σας είπα, συναντηθήκαμε τον πρόεδρο αυτού του Συμβουλίου και μας έδωσε και μία κατάσταση προτεραιοτήτων υπό τη σκοπιά βέβαια του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου. Πρώτος στόχος, πρώτη προτεραιότητα, απομάκρυνση του Καντάφη. Καμία συζήτηση μαζί του, καμία συζήτηση με την οικογένειά του. Δεύτερον, μα ζητούν να μεταφέρουμε το μήνυμα στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ζητούν μεγαλύτερη αναγνώριση του Εθνικού Συμβουλίου θεωρούν ότι πρέπει να αναγνωριστεί ω νόμιμη κυβέρνηση τη Λιβύης. Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη ομιλητέ που συναντήσαμε. Οι Λυβοί πρέπει να αναγνωρίσουν το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο. Τρίτον, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική προτεραιότητα από τον Ντελζαλή και ολου του αλλου συνομιλητέ που συναντήσαμε. Η Λιβύη πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Αυτή είναι η προτεραιότητά του Ήταν σαφές το μήνυμα, ηχηρό και το λάβαμε από όλους τους συνομιλητές εκεί. Όλους όσους ε, είδαμε, ε, όλοι όσους είδαμε, ζητούσαν ευρωπαϊκή υποστήριξη και το ζητούσαν έντονα. Είχαμε την εντύπωση ότι δεν το ζητούσαν, δεν ζητούσαν στήριξη οικονομική, χρηματική, διότι έχουν ε, την ε, εντύπωση και την επίγνωση, θα έλεγα, ότι είναι μια πλούσια χώρα, εύπορη χώρα. Και όταν ο πλούτος της χώρας αυτής θα είναι διαθέσιμος, θα μπορούν να πληρώσουν για οποιαδήποτε υπηρεσία. Τώρα όμως αυτό που χρειάζονται και αυτό που ζητούν είναι η υποστήριξή μας, τεχνική υποστήριξη. Και καταγράψαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτεραιότητες. Δημιουργία δυνατοτήτων και υποδομών, ηγεσία, ε, δεξιότητες διαχείρισης, στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των εξάρτητων μέσων ενημέρωσης, ρόλος μέσων ενημέρωσης, επικοινωνία. Ο ρόλος της επικοινωνίας τονίστηκε πάρα πολύ έντονα και υπήρχε και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Έχω και να σας δείξω κάτι. Να σας δείξω αν το βρω αν το έφερα, δεν το έφερα. Ήθελα να το φέρω και να σας το δείξω, αλλά την πρώτη εφημερίδα θέλω να σας δείξω. Sorry. <laughs> I, I did some presentation today. Έκανα κάποια παρουσία σήμερα, αλλά δυστυχώς άφησα το συγκεκριμένο φάκελο στο σπίτι. Ε, ή στο γραφείο μου τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν μια δισέλιδη εφημερίδα φοιτητική που με πολύ περηφάνεια μας την επέδειξαν οι φοιτητέ, την πρώτη ελεύθερη εφημερίδα της Βενγκάζης. Ζητούσαν λοιπόν στήριξη, στήριξη στα ανεξάρτητα μίντια, στην επικοινωνία, στην εσωτερική επικοινωνία μεταξύ του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου, της Κοινωνίας των Πολιτών, της Κοινωνίας των Πολιτών και του πολιτικού επίπεδου, αλλά και επικοινωνία από τη Λιβύη προς την Ευρώπη. Θέλουν δηλαδή εμείς να ενημερωθούμε, να μάθουμε ποια είναι η κατάστασή τους, τι επιθυμούν, τι προσδοκούν, ποια είναι η κατάσταση. Ασφάλεια τώρα. Μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το τόνισαν πάρα πολύ. Διαχείριση συνόρων. Δεν έχουν κανένα, ε, κανένα συνοριακό έλεγχο. Παιδεία, υγεία, οικονομία και δημοσιοοικονομικά, διαχείριση δημοσιοοικονομικών. Όπως βλέπετε υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος πάρα πολύ σημαντικών τομέων παρέμβασης. Εμείς αποκομίσαμε την εντύπωση ότι η στήριξη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να ξεκινήσει ευθύ αμέσω. Όταν λέω ευθύ αμέσω εννοώ σήμερα. Φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίφαση σε σχέση ή σε σύγκριση με τη ρευστότητα που υπάρχει, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες οι Λίβοι. Θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους και περιμένουν κυρίως από την Ευρώπη να τους υποστηρίξει αυτή την αλλαγή. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αφιερώσουμε όλες μας τις προσπάθειες για να διατηρηθεί αυτή η ορμή και αυτή η πολιτική βούληση των αναδυόμενων δημοκρατικών θεσμών. Μικρή είναι η διεθνής παρουσία τουλάχιστον μέχρι στιγμής και τουλάχιστον στη Βενγάζη. Ο συντονιστής ή το προσωπικό από τις Αδενωμένα Έθνη έφτασε μόλις προχθές στη Βενγάζη. Πάντως έφτασαν ή του ΟΗΕ εκεί και θα μπορέσουν να αναλάβουν ε, τα καθήκοντα του συντονισμού ή κάποια τέλο πάντων από τα καθήκοντα του συντονισμού ή της ανθρωπιστικής βοήθειας ή άλλες κάποιες δραστηριότητες ε, που αναλαμβάνει ο ΟΗΕ και σχεδιάζουν να πάνε και στην Τρίπολη. Αυτό το οποίο προτείνουμε και σήμερα το πρωί Μια αντίστοιχη αναφορά έκανα ε, στους 27 ε, πρέσβεις ε, γιατί έχει ζητηθεί να έχουμε παρουσία, ευρωπαϊκή τεχνική παρουσία στη Βενγκάζη, να ανοίξει ένα γραφείο εκεί, ώστε να στηριχθούν αυτές οι τεχνικές προσπάθειες, να γίνουν οι αναλύσεις που πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, ή πρωτοβουλία, πρωτοβουλίας, από τη στήριξη της, της κοινωνίας των πολιτών μέχρι την, τον έλεγχο των συνόρων. Ναι, υπάρχει μια καλή ανάλυση, μια καλή αξιολόγηση, καλή κατανόηση της κατάστασης. Και προς ενημέρωσή σας να σας πω ότι η σημερινή παρουσίαση που έκανα στους 27 πρέσβης Κόψ ήταν θετική. Όλοι τους ε, αντέδρασαν θετικά σε όλα αυτά τα σημεία δηλαδή και στην ιδέα του να ανοίξει ένα τεχνικό γραφείο εκεί. Και αυτό που μας ε, έδωσαν ως σύσταση σήμερα είναι να προσέξουμε να μην δώσουμε την εντύπωση ότι αναγνωρίζουμε μόνο το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο. Να δώσουμε όμως την εντύπωση ότι αναγνωρίζουμε γενικώ το κίνημα αυτό που ίσως θα είναι το μελλοντικό κίνημα στη Λιβύη. Δεν θέλουμε να δοθεί εντύπωση ότι θέλουμε να διαιρέσουμε τη Λιβύη. Δηλαδή ότι φτιάχνουμε κάτι στη Βενγάζη θέλουμε να την αποχωρήσουμε, να την αποσπάσουμε από την ε, Τρίπολη. Σίγουρα η Βεγγάζη μέχρι στιγμής είναι το μόνο μέρος όπου μπορούμε να κάνουμε κάτι με σχετική ασφάλεια. Αλλά είναι προφανές ότι όταν είναι ελεύθερη και η Τρίπολη, όταν είναι ανοιχτή η Τρίπολη, τότε αυτού του είδους ε, οι προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν και στην Τρίπολη. Θα μεταφέρουμε τις προσπάθειές μας δηλαδή ε, και φυσικά το επικεντρώμα θα είναι οι γυναίκες, οι νέοι, η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ζητούν την υποστήριξή μας. Πανερχόμενο στο πρώτο ερώτημα, γιατί είμαι στην ε, ΕΕ και τι κάνω εκεί. Η απάντηση καλύτερη μπορώ να σας δώσω είναι αυτή η διαπηρεσιακή αποστολή. Γιατί αυτό που λέει η λέξη ε, είναι ότι η υπηρεσία την οποία έχω την τιμή να, την οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, ε, έκανε αυτή την αποστολή. Ήταν πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα και ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι και εμείς γενικά και εγώ προσωπικά ούτε αλληλεπικάλυψη θέλουμε να κάνουμε ούτε να περιπλέξουμε τη ζωή των αρμόδιων για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΚΟ, η ΕΚΟ θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της. Δεν είμαι πολιτικός σύμβουλος ε, του γραφείου αυτού, ούτε ελεγκτής του γραφείου αυτού. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους του ΕΚΟ στη Βενγάζη, μας δίνουν ε, τη δική τους εικόνα, την ανάλυση της κατάστασης και συνεργαζόμαστε μαζί τους, βλέπουμε τι έχουν να μας προτείνουν, ε, ακούμε τις συστάσεις τους και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μαζί κάτι. Θέλουμε δηλαδή και τη φάση της επίγουσας βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας να τη συνδυάσουμε. Αυτά έχουμε κάνει λοιπόν στην αποστολή που σας περιέγραψα και στην ακτή λεφαντός τους προσεχείς ημέρες γιατί ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα πάμε εκεί, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο και εκεί. Κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουμε κάνει στην Βενγάζη και στη Λιβύη. Ευχαριστώ. Bien, Καλώς, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πολύ συγκεκριμένη και ζωντανή παρουσίαση. Πολλοί συνάδελφοι στον το λόγο θέλουν να αντιδράσουν. Η κυρία Χάνκης. Ευχαριστώ πολύ. Τα σχέδια τα οποία μας παρουσιάσετε θα είναι πάρα πολύ θετικά, πιστεύω, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τι επακριβώς γνώμη έχετε για το μέλλον. Ύστερα από αυτή την επαναστατική περίοδο, μετά το τέλος της επαναστάσεως, υπάρχουν πραγματικές βάσεις, ευκαιρία για δημοκρατία, σταθεροποίηση, των δημοκρατικών θεσμών. Δηλαδή, πώς μπορούμε εσείς, εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους βοηθήσουμε να αποφύγουν αυτή την ε, ταραγμένη περίοδο. Χωρίς να περιπέσουν σε σφάλματα. Τι γνώσεις έχετε εσείς. Οι δικές μου πληροφορίες βέβαια δεν αρκούν, αλλά βλέπω ότι το επαναστατικό κίνημα δεν ξέρω εγώ, αλλά είναι ας πούμε ενωμένο, είναι διαιρεμένο. Τι ευκαιρίες μπορεί να, τι ευκαιρία μπορεί να έχουν και ανάπτυξη ενός νέου καθεστώτος μετά. Ευχαριστώ Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Μιώτσο για αυτήν την πρώτη συζήτηση εδώ. Η έκθεση του μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μια πιο πολιτική συζήτηση στο πρώτο κομμάτι με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Παπόφσκη. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς μείναμε σε αυτά τα χωρισμένα κομμάτια της ημερήσιας διάταξης. Γιατί χωρίστηκε η ημερήσια διάταξη έτσι. έκθεση τώρα του κυρίου Μιάντσο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το να πάμε επί τόπου για να αντιληφθεί κανείς ποια είναι η κατάσταση, ε, για να δει συγκεκριμένα τι έχει γίνει σε σχέση με τις αρχικές εξελίξεις. Και νομίζω ότι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αυτό το ακριβώς το πρόβλημα, ότι δεν είχε εικόνα σαφή της κατάστασης. Δεν είναι ασαφής η εικόνα που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εντύπωση λοιπόν την οποία εσείς μας μεταφέρετε για την ε, το ότι δημοκρατική φύση αυτής της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική. Δεδομένου δε ότι το δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν στοιχεία εμφυλίου πολέμου, στοιχεία εξέλιξης προς τη δημοκρατία και ανάλογα με το τι θα επικρατήσει η απάντηση που δίνει κανείς είναι διαφορετική, γιατί δεν έχουμε μόνο δημοκρατική επανάσταση, έχουμε και εμφύλιο πόλεμο ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν ρωτώ, έχετε την εντύπωση αυτή ε, ότι πρόκειται για μια δημοκρατική επανάσταση και ε, μόνο για τη Βενγάζη ή γενικότερα ισχύει κατά την απόψή της στη χώρα. Ε, οι φίλες, οι φατρίες καλύτερα ε, επιτείνουν να επικρατήσουν ή είναι τα δημοκρατικά αιτήματα του λαού. Πώς βλέπετε και πώς κρίνετε τις εξελίξεις. Ως προς δε την φύση της συγκρούσεως αλλά και ως προς το ζήτημα το σχετικό με τα θύματα, με τη δυναμική, την εξέλιξη της υπόθεσης. Έχετε μπορέσει να καταλήξετε σε μια κάποια τάξη στην υπόθεση αυτή. Έχετε βάλει σε μια σειρά φερρυπίν τα αριθμητικά στοιχεία, τα στατιστικά, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και ε, δεν μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Έχετε βρει μια σειρά εκεί μέσα. αληθεύει ότι υπάρχει κάποια γραμμή στο μέτωπο που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει την ανάπτυξη μιας εκεχηρίας ή πάντως τη θεροποίηση κάπως της κατάστασης ή πώς βλέπετε εσείς το ενδεχόμενο μιας εκεχηρίας. Ο πρόεδρος Δανζοίδης έθεσε ένα ερώτημα σχετικό. Από την πρώτη σας εμπειρία λοιπόν, πώς ε, βλέπετε να προχωράει ο ρόλος ε, διαχείρισης της κρίσης στο πλαίσιο της, εξωτερικής, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ξέρω ότι σας ετέθη το ερώτημα, αλλά πώς, πώς βλέπετε εσείς το ρόλο σας. Ο κύριος Φάκερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τον τρόπο με τον οποίο, κύριε Μιώτσο, ε, ενημερώσατε την Επιτροπή μας και την προσωπική σας στράτευση στην υπόθεση αυτή. Βλέπουμε ότι προσπαθείτε να είστε στο δυνατόν πιο συγκεκριμένος. Έχω λοιπόν μια ερώτηση. για την κατάσταση στην Κυριναϊκά, στην Κυριναϊκή δηλαδή, ή την Τρίπολική, Τριπολιτική, που μας αναφέρατε και εσείς. Και βεβαίως, εάν ο κόσμος τη Βενγάζη θέλει να παραμείνει η Λιβύη ως ενιαίο κράτος, να διαφυλαχθεί δηλαδή η ενότητα του κράτους, πιστεύετε ότι θα πρέπει να δούμε και τι λένε οι άλλοι, η άλλη πλευρά τι λέει δηλαδή όταν συνομιλείτε μαζί τους. Έχουν επαφές με κάποιους ομοειδεάτες ενδεχομένως στην, στην Τρίπολη της Λιβύης όπου ε, ενδεχομένω ακόμη δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, να εκφράσουν την ελεύθερη βούλησή τους. Γιατί η Τρίπολη μας δίνει μόνο εικόνες προπαγάνδας. Και ίσως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν τον εκδημοκρατισμό, που θέλουν να απαλλαγούν από τον Καντάφη, ίσως δεν είναι σε θέση να εκφράσουν την ελεύθερη βούλησή τους. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες επαφές, κάποιοι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων εκεί. Τρίπολης δηλαδή και Βενγάζης. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη. Ο κόσμος τι λέει. Γιατί από τις ε, αναφορές του τύπου τουλάχιστον βλέπουμε δρόμους που αναπτύσσονται εχθροπραξίες, ανεβαίνουν οι μεν, κατεβαίνουν οι δε. Τι λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια κατάσταση εμπόλεμη τελευταία ανάλυση. Πόσο θα αντέξουν ακόμη να πολεμάνε. Γιατί είναι προφανές ότι η άλλη πλευρά έχει καλύτερο εξοπλισμό. Έχουν βαρύ εξοπλισμό, βαρύ οπλισμό που δεν διαθέτουν οι άλλοι. Επομένως τι μπορούμε να κάνουμε και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε αυτούς τους ε, επαναστάτες, τους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε ακόμη και εξοπλισμό, Φερρυπίν. Οπλισμό ώστε να μπορούν να πολεμούν ίσης ώρες επίσης ώρες με το καθεστώς του Καντάφη. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Και τελευταία μου ερώτηση. Πώς αισθάνεστε εσείς που θα εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ξέρετε ότι είναι πολύ αντιφατικές οι θέσεις που εκφράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ την εμπλοκή μα στη Λιβύη. Υπάρχουν υπουργοί όπω ο δικό μου που καθημερινά επαναλαμβάνουν πως δεν σκοπεύουν να συμμετάσχουν ε, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τι μπορείτε να μας μεταφέρετε λοιπόν εσείς ε, από την εικόνα που έχετε για αυτή την κατάσταση. Αυτή η απουσία ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την κρίση στη Λιβύη. Ευχαριστώ κυρία Λόσινγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούγονται πολλές φορές ε, παράπονα διαμαρτυρίες ότι έχουμε χωρίσει τη Λιβύα και τη U4 σε δύο διαφορετικά θέματα μέρη τη ένταξη. Δεν θα το αναπτύξω και εγώ. Απλώς επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να σας ρωτήσω για τη U4. Γιατί είδα, διάβασα με προσοχή την βιογραφία σας, το βιογραφικό σας. Βλέπω ότι είστε και γιατρός, έχετε καταπληκτικές γνώσεις και ικανότητες, έχετε εμπειρία πολλαπλή από ανάπτυξη επιχειρήσεων για κατάσταση ανθρωπιστική ανάγκης, όχι ιατρική, ανθρωπιστική. Ε, και σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα να σας διατυπώσω την ερώτηση, γιατί πριν από λίγο σήμερα είχαμε τη συζήτηση της UFOR εδώ. Την κατάσταση λοιπόν εσείς στη Λιβύη πώς την βλέπετε. Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη ανθρωπιστικών μέτρων, μέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανθρωπιστική βοήθεια εν προκειμένου, ενώ η ιατροφαρμακευτική βοήθεια, ε, επισητιστική βοήθεια. Αυτό θέλω να ακούσω από σας Πώς βλέπετε από τη δική σας τη σκοπιά την κατάσταση, ξέρω ότι είστε πολύ έμπειρος, στην υπόθεση αυτή της αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών κρίσεων χρειάζονται ιατροφαρμακευτική βοήθεια ή άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με στρατιωτική βέβαια προστασία. Και ένα άλλο ζήτημα για τους ε, πρόσφυγες που δεν συζητήσαμε αρκετά σήμερα γιατί ακούστηκαν πολλά για μέτρα βοήθειας ανθρωπιστικής στη Λιβύη, Μιλήσατε για τεχνική στήριξη και ούτω καθεξής. Αλλά μεγάλο καθήκον ανθρωπιστικό είναι αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται στα σύνορα της Αιγύπτου, ουσιαστικά εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να τους φέρει φαΐ, κάποιος να τους φέρει νερό. Και πρέπει να υπάρξει και η συνοδεία στρατιωτική που θα διασφαλίσει την πρόοδο αυτών των ανθρωπιστικών ε, μέτρων. Ερωτώ λοιπόν, από τα όσα μας είπατε καλά κατάλαβα ότι εστίαση δίνεται περισσότερο στην ανάπτυξη της κοινωνίας των, πολιών, των πολιτών, τη βοήθεια των δημοκρατικών, προς τις δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά λιγότερο προς τα ανθρωπιστικά και μιλήσατε και για βοήθεια στον έλεγχο των συνόρων. Είπατε ότι υπάρχει έλλειμμα αυτή τη στιγμή στον έλεγχο των συνόρων. Πώς το βλέπετε λοιπόν αυτό. Θα μπορούσε ενδεχομένω η Frontex να αναλάβει μια ενισχυμένη δραστηριότητα εκεί και η U4 υπό όρους θα μπορούσε ενδεχομένω να στηρίξει τις δραστηριότητες Frontex εκεί. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βιώτσο για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω παρακολουθήσει το θέμα της Λιβύης ως ηγήτρια για τη Συμφωνία πλαίσιο τους τελευταίους μήνες και οφείλω να πω ότι δεν με εκπλήσουν τα όσα ακούω. Αυτά που μας είπατε ήταν για μένα αναμενόμενα από όσα έχω δει μέχρι τώρα στην Τρίπολη και τη Βενγάζη και από όσο έχω εγώ αναλύσει την κατάσταση με βάση πληροφορίες που λαμβάνουμε. Με ενθαρρύνουν μάλλον αυτά που λέτε. Δεν με αποθαρρύνουν, δεν με εκπλήσουν πάνω απ' όλα. Και είναι πολύ σημαντικό πιστεύω το ότι οι άνθρωποι με του οποίου έχετε συνομιλήσει ζητούν τέτοιου είδου βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε η ώρα να του την προσφέρουμε την ε, στήριξη αυτή, να του βοηθήσουμε να ετοιμάσουν το μέλλον του. Ο Καντάφη ανοίξει το παρελθόν. Μπορεί να είναι ακόμα εκεί, αλλά ανοίξει το παρελθόν. Τέλειωσε αυτό. Έχει λήξει. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε πια μαζί του. Δεν ελέγχει πια τη χώρα, κυρία Λέσσινγκ, δεν ακούγεται δυστυχώ. Πρέπει επομένως να οικοδομήσουμε το μέλλον. Και αυτό μαζί με εκείνους που ήδη είναι και θα αποτελέσουν την ε, βριακή μορφή ε, της μελλοντικής εξουσίας στη Λιβύη. Άρα είναι καλό το ότι αναγνωρίζουν πως δεν επαρκούν από μόνες τους οι δυνάμεις τους και ζητούν ε, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη ικανότητων, για capacity building δηλαδή. Και όπως είπα, ε, και εμένα αυτό ακριβώς, ε, έχω αυτή, ακριβώς την εντύπωση είχα, ιδιαίτερα στην επίσκεψη στη Βενγάζη, ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, όπως ξέρετε. Με την κυρία Φερέρο Βάλτνερ είχαμε, είχαμε ξεκινήσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των ε, νοσοκόμων ε, και του γιατρού από την Παλαιστίνη, των βουλγαρίδων ε, νοσοκόμων και του γιατρού από την Παλαιστίνη και βέβαια το μεγάλο αγώνα για την καταπολέμηση του ιού του AIDS στη Βενγκάζη μας είχε καταπλήξει θερμότατη υποδοχή που μας επιφύλαξαν οι γιατροί και οι νοσοκόμες, όλοι οι γιατροί και νοσοκόμες στη Βενγκάζη, Η, η στήριξη και η αναγνώριση της ε, η προσπάθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα που είχε τεράστια σημασία για αυτούς, και κρίσιμη σημασία και που είχε τεράστια απήχηση στην Βεγγάζη και έκανε τεράστια έφερε τεράστιες αλλαγές διότι άλλαξε από το 2008 από εκείνη την ώρα που εμείς βοηθήσαμε για τον αγώνα κατά του AIDS ε, ε, άλλαξαν πάρα πολλά το, από το 2008 αμέσως για αυτούς τους 300 τόσους που είχαν εμολυνθεί από τον ιό του AIDS, γενικά στην πρόληψη. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ, πολλά να προσφέρουμε και πρέπει να πω ότι εκείνη την εποχή ήταν και πολύ ε, διστακτική, δεν τορμούσαν να μιλήσουν ανοιχτά. Είχα μιλήσει με μια γιατρίνα εκεί που ήταν ε, κάπως πιο μιλητική θα έλεγα, το μεσημέρι τρώγοντας μαζί της, κατηδίαν, τη ρώτησα τι βλέπει ως πραγματική αιτία της επιδημίας του HIV-AIDS. Και απάντησε δεν μπορώ να εμπλακώ σε πολιτική συζήτηση. Πολύ χαρακτηριστική απάντηση. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να απαντήσουμε, να ανταποκριθούμε σε αυτά τα αιτήματα ως προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω 100% με την ιδέα της παρουσίας μας εκεί. Νομίζω ότι είναι σύμφωνο και με το ψήφισμα που έχουμε ήδη εγκρίνει. Όταν μιλούμε για την ανάπτυξη επαφών, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αναγνώριση πολιτική κάποιων συγκεκριμένων τάσεων. Υπάρχει αναγνώριση ότι υπάρχει μία οντότης λιδική που ίσως αποτελέσει και το μελλοντικό ε, μόρφωμα της κυβέρνησης της Λιβύης και πρέπει να τη βοηθήσουμε να αναπτύξει το δυναμικό εκείνο, το, το, τις ικανότητες εκείνες που θα, θα έχουν κρίσιμη σημασία για την, για την εξέλιξη αυτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και θα ήθελα και να σας ενθαρρύνω βέβαια στη γραμμή αυτή, δηλαδή να ε, αναπτύξετε εκεί την παρουσία μας. Με ιδιαίτερη να όμως να μην θεωρηθεί αυτό ότι έχει σαν αποτέλεσμα τη διχοτόμηση της Λιβύης και εν προκειμένου, θα ε, ήθελα να ρωτήσω ερωτήσεις πολύ σημαντικές που έχουν κάνει και ο κύριος Πάσκου βέβαια και ο κύριος Γουαλτιέρη με βρίσκουν συμφωνεί, αλλά θα ήθελα να προσθέσω. Τι νόημα έχει αυτή η ανθρωπιστική επιχείρηση που έχει υποσυζήτηση το Συμβούλιο θεωρητικά αλλά δεν γίνεται τελικά τίποτα γιατί ε, αποφεύγουν την διατύπωση του συγκεκριμένου αιτήματο. Εσείς μας λέτε ότι αυτό ακριβώς χρειάζεται ίσως όχι τόσο πολύ ανθρωπιστική ε, στήριξη, ίσως ιατροφαρμακευτική βέβαια, ναι, αλλά περισσότερο χρειάζονται από ό,τι φαίνεται οικοδόμηση δυνατοτήτων, capacity building, σε αυτό θέλουν στήριξη. Άρα, ε, σε ποιο βαθμό συμπίπτουν αυτά που βλέπετε σε αυτή τη Βενγάζη και αυτά που συζητούνται εδώ στις Βρυξέλλες. Και επίσης, Ε, υπήρξαν αιτήματα για οπλισμό Φερρυπίν. Χωρίς να λέω ότι θα υποστήριζα ένα τέτοιο αίτημα, αλλά, γιατί δεν το υποστηρίζω, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν σε έχουν ζητήσει ή αν έχουν ζητήσει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή του καθεστώτος του αποκλεισμού όπλων του εμπάρκου δηλαδή στο καθεστώς του Καντάφη και όχι μόνο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά από τον Νότο ιδιαίτερο, γιατί από εκεί προέρχονται προ Αυτά νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με την τελευταία παρέμβαση της ε, Άννα Γκόμες, μήπως μπορείτε να μας διευκρινίσετε περισσότερα σε σχέση με τα αιτήματα των, ε, που ακούσατε στη Βενγάζη και σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει στη δυτική πλευρά ε, σε ζώνες ε, στις οποίες ε, συνεχίζεται η, συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Για, πολύ πιο συγκεκριμένα μιλάω για τη Μιστράτα. Επειδή μιλήσατε συγκεκριμένα για την Βενγάζη και για ένα ανατολικό κομμάτι που είναι από ό,τι κατάλαβα σχετικώς ασφαλές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. κατά, πόσο, κατά πόσο είχαμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια βάση για εκδημοκρατισμό. Ναι, σαφέστατα. Συναντήσαμε κόσμο μόνο στη Βενγάζη ε, από διάφορα επίπεδα, νέους, ακαδημαϊκούς, δασκάλους, πολιτικούς, γυναίκες. Συναντήσαμε λοιπόν ε, ένα ευρύ φάσμα ε, πολιτών, πολιτικούς από το Μεταβατικό Συμβούλιο, ε, τον επικεφαλής της ασφάλειας της αστυνομίας και έχουμε μια πραγματική αίσθηση ότι υπάρχει βάση για δημοκρατία οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους ε, συνομιλήσαμε, θα προσπαθήσω να πάω λίγο πιο πίσω να σας εξηγήσω γιατί, τι θέλω να πω. Είδα καταπληκτικούς ανθρώπους μετά από 42 χρόνια να λένε για πρώτη φορά στη ζωή μας είμαστε περήφανοι για τη σημαία μας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε λίδοι. Είμαστε περήφανοι που γράφουμε ένα σύνταγμα. Πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν το άκουσα αυτό. Νέοι άνθρωποι να λένε ότι χαιρόμαστε τόσο πολύ και είμαστε περήφανοι που γράφουμε ένα σύνταγμα. Θα ήθελα και εγώ ε, να ε, να ακούσω τα παιδιά μου να λένε ε, ότι, θα, ότι είναι περήφανα για το σύνταγμά μας, ε, ότι είναι περήφανα για το σύνταγμά τους και τη σημαία τους, ενδεχομένως να μην ξέρουν καν τι γράφει το σύνταγμα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι μπορούν να συμμεριστούν αυτό το συνέστημα που σας περιγράφω. Και γιατί λέω ότι είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει βάση για δημοκρατία. Πολλοί ε, από όσους ε, γνωρίσαμε ε, μας είπαν ότι το θέμα των φυλών δεν είναι πραγματικός λόγος, ούτε η θρησκεία είναι ο πραγματικός λόγος για την, πραγματική, για την επανάστατη για την Επανάσταση. Το θέμα που, λέει, το θέμα που αναφέρεται συνεχώς ε, σε σχέση με τις φυλές και τη θρησκεία είναι ε, κάτι που έχει εφεύρει ο Καντάφη ο ίδιος. Για μας δεν είναι ένα πραγματικό ζήτημα αυτό. Αυτό λένε οι άνθρωποι επί τόπου. Είμαστε μουσουλμάνοι, λένε οι ίδιοι. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μουσουλμάνοι. Αλλά για μα το να είμαστε μουσουλμάνοι είναι όπω είστε εσεί χριστιανοί. Είμαστε κατά τη Αλκάιντα, είμαστε κατά ε, το, των εξτρεμιστικών στοιχείων. Κατά πόσο υπάρχει τώρα πραγματική ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι, σε, σε μερικές περιοχές υπάρχει. Στη Μισράτα, για παράδειγμα, χρειάζονται ε, κάποια βασικά αγαθά. Χρειάζονται τρόφιμα, χρειάζονται ε, φάρμακα. Είδαμε την ICRC, είδαμε τον Γαλλικό Ρήτρο Σταυρό, είδαμε πολλούς φορούς που προσπαθούν να βοηθήσουν. Υπάρχει μια πραγματική ανάγκη προετοιμασίας ε, μιας ανθρωπιστικής βοήθειας. Για την ώρα περιμένουμε, αλλά η αίσθηση που είχα εγώ, η εντύπωση που δημιουργήθηκε στην τελευταία μου αυτή επίσκεψη, αλλά και στις πρώτες δύο επισκέψεις που έκανα στη Λιβύη, και συμφωνώ με την κυρία Γκόμες όταν λέει ότι έχει παρέλθει ο Κατάφη. Ναι, ναι, Όντω, στο μυαλό των ανθρώπων έχει περάσει η εποχή Κατάφη, δεν τον θέλουν καθόλου, όμως εξακολουθεί να είναι εκεί και είναι ακόμη πάρα πολύ ισχυρό. μπορεί να έχει αλλάξει η στρατιωστική του τακτική, μπορεί να... Ε, μπορεί να κινηθεί στρατιωτικά πάρα πολύ γρήγορα. Οι αλλαγές είναι πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα χρησιμοποιούν ε, άλλα οχήματα και πηγαίνουν από τη μία πόλη στην άλλη με δύο, σε δύο ώρες. Αν δηλαδή 44-4x4 ε, και βαρέα όπλα ε, είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσει κανείς στη Βεγγάζη. Συνεπώς, δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος έλεγχος από την ε, ζώνη απαγόρευσης πτήσεως. Υπάρχει πρόβλημα με τον έλεγχο τέτοιου είδους μετακινήσεων. Άρα η κατάσταση είναι ακόμη πάρα πολύ ρευστή και χρειαζόμαστε να έχουμε στο μυαλό μας αυτή την ενδεχόμενη στρατιωτική παρέμβαση για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής κατάστασης για την ώρα νομίζουμε ότι δεν χρειαζόταν. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όταν θα χρειαστεί. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε τώρα, να προετοιμαστούμε, γιατί η κατάσταση για την ώρα είναι ακόμη πάρα πολύ ρευστή και πάρα πολύ εύθραυστα όλα. Πραγματικά αυτή είναι η εντύπωση όχι μόνο η δική μου, αλλά και όσων βρίσκονται εκεί. Όσον αφορά τη Μισράτα και κάποιες άλλες ε, ε, μικρές πόλεις όπου, υπάρχουν, όπου γίνεται ο πόλεμος. Ναι, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θέλω να το, επαναλάβω αυτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Μέχρι τώρα αξιολογούσαμε την κρίση της Λιβύης ε, όχι μόνο βάσει των όσων ακούγαμε στο CNN, στο BBC και ε, βάσει των επισήμων ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, εν πάση περιπτώσει. Βλέπαμε για παράδειγμα τη φωτογραφία μέσω δορυφόρου από τη Μισράτα, από την Τρίπολη, από εδώ, από εκεί. Δεν έχουμε τα μάτια μας εμείς εκεί επί να βλέπουμε τι γίνεται. Ούτε το CNN, ούτε η Al Jazeera καν. Ε, παίρνουν πληροφορίες και εικόνες ε, στις εμπόλεμες ζώνες όπου διαδραματίζονται οι μάχες ε, είναι ε, εικόνες που έχουν πάρει από άλλους. Πριν από δύο μέρες η ICRCP μπόρεσε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πει. Η Τρίπολη. Γνωρίζουμε ότι η Τρίπολη έχει μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό το πρόβλημα, δεν είναι κρίσιμη η ανθρωπιστική κατάσταση, όμως όλος ο κόσμος πραγματικά φοβάται να ανοίξει το στόμα του. Όταν πήγαμε στην, Τρίπη, πριν, στην Τρίπολη πριν από ένα μήνα, γνώρισα Ευρωπαίους διπλωμάτες, Ευρωπαίους πρέσβεις ε, της Ιταλικής αποστολής. Ήταν μια εσωτερική συζήτηση με πρέσβεις και διπλωμάτες. Φοβόντουσαν να ανοίξουν το στόμα τους για τις συνθήκες που επικρατούν εκτός της Ιταλικής πρεσβείας. Αυτή ήταν η δική μου εντύπωση. Ο Ιταλός πρέσβης φοβόταν να μας πει ειλικρινά πώς ήταν τα πράγματα σε μια εσωτερική συνάντηση της Ιταλικής αποστολής, της Ιταλικής αντιπροσωπείας. Τώρα, πώς η Τινησία ή η Αίγυπτος μπορεί να αντιδράσει. Για την ώρα δεν ε, Εμείς η επιχείρηση που έχουμε ε, μέχρι τώρα δρομολογήσει, χάρη στην ΕΚΟ και χάρη σε άλλους φορείς, ήταν ε, πάρα πολύ καλή. Αν θυμάμαι περίπου χίλια άτομα έχουν φύγει από την περιοχή, έχουν φύγει από τη Λιβύη και έχουν πάει στην Τινησία ή στην Αίγυπτο. Για την ώρα, στα σύνορα με την Αίγυπτο υπάρχουν όχι πάνω από 2.000, 1.500, άτομα Αφρικανοί που περιμένουν να μεταφερθούν στις χώρες τους. Ε, γιατί η Αίγυπτος δεν τους επιτρέπει να μπουν ε, στο, στην Αιγυπτιακή επικράτεια. Και ε, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσπαθεί να οργανώσει την επιστροφή του στην Γκάνα, στο Τσάντ, ε, ε, σε πολλές χώρες της Νότιας Αφρικής ε, και όχι στο Μπαγκλαντές, στην Απονατολή, στις Φιλιππίνες. Η ανθρωπιστική κατάσταση στα σύνορα για την ώρα ελέγχεται και οι Αιγυπτιακές αρχές και οι αρχές της Τινησίας ε, συνεργάζονται πάρα πολύ καλά, επιτρέπουν ε, τους, τις ανθρωπιστικές δυνάμεις να περάσουν τα σύνορα και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ε, ώστε να περιπλέκεται η, η ζωή όσων προσπαθούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα, όσον αφορά την υποστήριξη, να σας πω την αλήθεια, εμένα δεν μου ζήτησε κανείς όπλα. Αλλά μας έχουν πει ναι, πρέπει να μας υποστηρίξετε με όσο το δυνατόν, ε, ε, με όλους τους, τους τρόπους ε, με όλους τους δυνατούς τρόπους και στη Μισράτα και σε άλλες πόλεις. είναι πολύ σαφές το μήνυμα που προσπάθησαν να στείλουν χωρίς να αναφέρουν καν τα όπλα. Οπότε, όσον αφορά τώρα το θέμα της Απόκληση απόψεων, διάσταση απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώ, λέω εγώ ευτυχώ, δεν έχουν καταλάβει ότι εμείς μεταξύ μας διαφωνούμε. Εμένα με βλέπαν ως Ευρωπαίο αντιπρόσωπο και έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Δεν κάνουν τώρα πολύ τη διάκριση ποιοι διαφωνούν, ποιοι συμφωνούν, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση είναι και πάλι πραγματικά πάρα πολύ ρευστή. Και από ψυχολογικής απόψεως αυτή τη στιγμή ε, μπορεί να είναι υπέρ μα, αλλά αύριο μπορεί να μας καταδικάσουν άμα, άμα εμείς ε, σταματήσουμε ένα πλοίο που πηγαίνει όπλα στη Μισράτα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερο να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να, να δώσουμε την απάντηση που ε, η κοινή γνώμη περιμένει από την Ευρώπη. Τουλάχιστον την απόδειξη ότι η Ευρώπη είναι εκεί. Θέλουν να αισθανθούν την παρουσία μας. Θέλουν νιώθουν ε, καλύτερα όταν βλέπουν ε, την Ευρωπαϊκή Σημαία και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόντα ε, στη Λιβύη. Αυτή είναι η πρώτη ελεύθερη εφημερίδα, τη Βρήκα, που δημοσιεύτηκε στη Βεγγάζη. έκλεγαν. Είναι μια απλή εφημερίδα και ήταν πάρα πολύ περήφανη για αυτή την πρώτη ελεύθερη ε, ε, εφημερίδα στην Κυριναϊκή και ε, ενδεχομένως και στη ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, όσον αφορά τη Frontex, τα αιτήματα για την υποστήριξη των ελέγχων στα σύνορα είναι πάρα πολύ ε, σημαντική πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ιδρύσουμε τελωνία. Δεν έχουν τελωνία. Αν περάσετε τα σύνορα, για παράδειγμα, προς την Αίγυπτο, υπάρχει ένα τελωνιακό σύστημα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρει τι μπαίνει κάποιο στη Λιβύη, α πούμε, κανένα δεν σου ζητάει τίποτα. Από πού έρχεσαι, τι θα κάνει, ε, αν έχει διαβατήριο, αν έχει θεώρηση. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να αναδιοργανώσουν το σύστημα τελωνίων του. Και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις της Frontex. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η ανάπτυξη των τελωνίων σε ε, πολιτικό επίπεδο τώρα, εντάξει δεν είναι ερώτηση αυτή, αλλά θέλω να σας δώσω μια ε, πληροφορία σχετικά. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν ε, η εντύπωση που αποκομίσαμε σε σχέση με όλους όσους έφυγαν από τη χώρα και κατά πόσο θα γυρίσουν όταν τελειώσει αυτή η κατάσταση, όταν τελειώσει ο πόλεμος. Εμείς ρωτήσαμε τι πιστεύετε για αυτούς τους μισό εκατομμύριο ανθρώπους που έφυγαν ε, και είχαμε την εντύπωση ότι ανησυχούν πάρα πολύ. Ότι ανησυχούν πάρα πολύ για όσους θα επιστρέψουν για την επιστροφή ενός μεγάλου αριθμού κυρίως Αφρικανών φτωχών ανθρώπων. Γιατί οι περισσότεροι ε, Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι τους, τους είχε προσλάβει ο ίδιος ο Καντάφη να κάνουν ε, δουλειές ε, με, με μισθό ψίχουλα και φοβόνται τι θα γίνει με την επιστροφή των ανθρώπων αυτών. Γιατί θα ήθελαν να ελέγξουν και να περιορίσουν όσο το δυνατόν ε, την επανεισρωή ε, αλλοδαπών στην ε, Λιβύη. Δεν ξέρω αν ξέχασα καμιά ερώτηση. Ενδεχομένως κάποια να ξέχασα. Ευχαριστώ να απαντήσω αν κάτι ξέχασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας ε, δώσατε μία περιγραφή της κατάστασης από πρώτο χέρι. Ήταν πολύ χρήσιμο για μας Επαναλαμβάνω, καλό θα ήταν βέβαια να είναι όλοι ε, οι υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική παρόντε ταυτόχρονα και ελπίζω σύντομα να γίνει αυτό, να έχουμε δηλαδή μια κοινή παρουσία για να έχουμε όλε τι ε, απαραίτητε πληροφορίε. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί και για τις επόμενες εβδομάδες ε, θα το παρακολουθούμε και το σύνεγγις και βέβαια Ελπίζω να είσαστε διαθέσιμος και στο μέλλον να έρθετε εδώ να μας κάνετε έτσι μια ενημέρωση για να έχουμε καλύτερη εικόνα για την κατάσταση επιτόπου. Η επιχειρησιακή προσφορά, αν θέλετε, που έχετε, η συνεισφορά σας θα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ολοκληρώσουμε την ε, απόψηνή μας συνεδρίαση με ένα διαφορετικό θέμα. Η υποεπιτροπή μας πρέπει να γνωμοδοτήσει ησυχία. Η υποεπιτροπή μας πρέπει να γνωμοδοτήσει για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με θέμα την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κυρία Χάνκης, που είναι εδώ, είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης αυτής. Να σας κάνω μια τεχνική υπενθύμηση. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 3 Μαΐου. Στην ΑΦΕΤ 25 Μαΐου θα εγκριθεί η έκθεση. Η έκθεση μάλλον, ε, θα πάει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Αυτές είναι οι ημερομηνίε. Κύριε Χάνκη, σας δίνω το λόγο. Παρουσιάστε τη γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ. Να σα κάνω κάποια σχόλια για το υπόβαθρο της γνωμοδότηση. Βάση της γνωμοδότηση ήταν η ανακοίνωση της Κομισιόν για την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπήρξαν κάποιες ε, συστάσεις ε, που θέλαμε να συμπεριλάβουμε από τη δική μας πλευρά, ως και ό,τι για την αντιτρομοκρατική πολιτική στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που είναι καθήλια αρμόδια, εγώ επικεντρώθηκα κυρίως στις πτυχές της ανακοίνωσης της Κομισιόν Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τον προπολογισμό τον αντιτρομοκρατικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο θεσμικό πλαίσιο, τις δομές, τις λειτουργίες πίσω από το μέτρο αυτό. Και είναι σαφές ότι ίσως δεν είναι θέματα της αρμοδιότητας της δικής μας υποεπιτροπής, αλλά η έκθεση της ΕΛΙΠΕ παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική γωνία. Εγώ θα τονίσω, όχι εδώ αλλά στη ΛΥΜΠΕ, ως και εισηγήτρια κάποια θέματα, γιατί δεν νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή μας ε, ε, μπορούμε να τα σχολιάσουμε, δεν είναι στο αντικείμενό μας. Αλλά να πω λίγα λόγια παρόλα αυτά. Εγώ προσωπικά έχω πολλές αμφιβολίες με την έκθεση της κυρίας Σίντβελτ. Δεν βλέπω κατά πόσον ε, μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί χωρίς να γίνει δεκτός ε, ένας, ένα μεγάλο επίπεδο κινδύνου. Η έκθεση της κυρίας Ινβέλτ μιλά για την παρακολούθηση της λειτουργίας της αντιτρομοκρατικής πολιτικής επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο ανεδαφικά τα όσα λέγονται στην έκθεση. Εγώ θα πρότεινα οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ένωσης αλλά και οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες δεν νομίζω ότι θέλουν να δώσουν αυτές τις πολύ λεπτές ευαίσθητες πληροφορίες δεν θέλω να τι κάνουν δημόσιες αυτές τι πληροφορίες. Ξέρω ότι μπορεί να μην συμφωνούν οι συνάδελφοι. Καταλαβαίνω βέβαια τις απόψει τους και τις διαφωνίε τους. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα τόσο μεγάλο επίπεδο κινδύνου. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Πιο ρεαλιστικό είναι να γίνει λοιπόν λόγος μόνο για την ανακοίνωση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την αντιτρομοκρατική πολιτική στο πλαίσιο της Επιτροπής μας και να μην μιλήσουμε για την έκθεση της κυρίας Ιντβέλτ. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Έχω κάποια ε, στοιχεία γνωμοδότησης ε, που θα σας τα διαβιβάσω ε, και πολύ σύντομα μπορώ να κάνω προφορικά μια συνόψηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι παγκόσμιο ο χαρακτήρα τη ε, τρομοκρατία, δηλαδή δεν ε, γνωρίζει σύνορα χώρε. Γι' αυτό θα πρέπει και η τρομοκρατική πολιτική να δώσει μια συνολική, μια παγκόσμια απάντηση. Η βάση δεδομένων στρατιωτικών πληροφοριών και ο Οργανισμό Άμυνα Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντε. Θα ήθελα να πω ότι τι τελευταίε εβδομάδε είχα την ευκαιρία να συζητήσω με ορισμένου επικεφαλεί ε, των εθνικών ε, μυστικών υπηρεσιών για μια κρόαση που οργανώσαμε και μας είπαν όλοι ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η στρατιωτική ενημέρωση, αυτές οι στρατιωτικές πληροφορίε, όχι η εσωτερική ε, πληροφορία για την εσωτερική ασφάλεια, γενικότερα. Τα δίκτυα εξωτερική ασφάλεια αλλά να προσθέσουμε και τις στρατιωτικές πληροφορίες στα καθήκοντα της αντιτρομοκρατικής δράσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω. Δεύτερον, προκειμένου να διευκολύνουμε τις κοινέ και παγκόσμιες δράσεις, οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εναρμονιστούν. Πρέπει να οριστούν οι όροι συνεργασίας και εγώ πιστεύω ότι πιο ξεκάθαρα θα πρέπει να γίνει διάκριση καθηκόντων και επιμερισμό των καθηκόντων μεταξύ της ε, κοινοτική υπηρεσίας και των εξωτερικών εθνικών υπηρεσιών. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά τα πράγματα, αυτός ο επιμερισμό καθηκόντων δεν είναι ξεκάθαρος. Δεν βλέπουμε ξεκάθαρα τις μορφέ συνεργασία, τη δομή τη συνεργασία. Και αν συμφωνήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο μηχανισμός συνένωση των προσπαθειών, αυτό το πρόβλημα πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή τη σχέση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής ε, ασφάλειας, δηλαδή οργανισμού και εξωτερικών υπηρεσιών. Επίσης, Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ε, των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η FTP και άλλα. Θα τα βρείτε και στην γραπτή μου νομοδότηση. Και θα πρέπει η αντιτρομοκρατική προσπάθεια να είναι σημαντικό στοιχείο των σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε, στα λεγόμενα failing states, σε κράτη παρείες, κράτη που έχουν αποτύχει και να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά στις προσπάθειές τους. Ένα ακόμη σημείο, η συνεργασία σε θέματα τη αντιτρομοκρατίας, σε συνεργασία και με τα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να επιταχυνθεί. Και προτεραιότητα των σχέσεων είναι κάτι που τονίζουμε στην έκθεση. Επόμενο σημείο, θέλω να τονίσουμε την όλο και αυξανόμενη διασύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονη αυτή η σχέση και η διασύνδεση σε πολλούς τομείς ε, και περιοχές. Ε, το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί και τη βασική πηγή χρηματοδότησης ε, των τρομοκρατών. Άρα μπορούμε αυτά να τα δούμε από κοινού. Διεθνές οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε νέες δομές για το νέο αυτό φαινόμενο. Έξω και πρέπει να τονίσουμε και τον, ε, τη σημασία της αξιολόγησης των απειλών, threat assessment. Θα πρέπει και να κάνουμε επίσης ανάλυση των τάσεων. Γιατί αλλάζουν οι τάσεις, ε, αλλάζουν οι μορφές των απειλών, ε, ε, το βλέπει κανείς αυτό ε, στην καθημερινότητα. Άρα και οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές θα πρέπει να έχουν αυτή την πολύ βαθιά ανάλυση τάσεων πρέπει να δούμε, ας πούμε, τη διαφοροποίηση της τρομοκρατίας, την στράτευση, στρατολόγηση μέσω ίντερνετ για παράδειγμα. Και ένα τρίτο Πολύ σπάνια γίνεται λόγο γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και στο μέλλον θα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο ίσως ε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, πώς μέσω δηλαδή μη κυβερνητικών οργανώσεων μπορούν να χρηματοδοτηθεί η τρομοκρατία. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Μπορείτε να τα διαβάσετε στη γνωμοδότησή μου. Και τώρα, κάτι πρακτικό. Κατάθεση τροπολογιών. 3η Μαΐου. Έχω ένα πρόβλημα όμως. Σε ό,τι αφορά την υποβολή και την έγκριση της έκθεσης για τις 24 Μαΐου. Επειδή είμαι μέλος της αντιπροσωπής με το Ισραήλ, είχα δεχθεί μια πρόσκληση για ε, να πάω ε, στην Κνέσετ, στην ε, Βουλή του Ισραήλ εκείνες τις ημέρες. Δεν θα είμαι παρούσα κατά την ε, ψηφοφορία. Θα είμαι στην Ιερουσαλήμ εκείνες τις ημέρες, μάλλον λαμβάνω. Ίσως θα μπορούσα να αναθέσω το καθήκον σε κάποιο άλλο μέλος του ΕΛΚ. Δεν ξέρω ακριβώς τι δυνατότητες υπάρχουν αλλά είχε προηγηθεί η αποδοχή της πολύ ευγενούς αυτής πρόσκλησης της Κνέσετ και δεν θα ήθελα να την αρνηθώ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα χρονοδιαγράμματος, η έγκριση είναι 25 Μαΐου στην ΑΦΕΤ. Θα είναι σημαντικό ούτως ή άλλως ε, να έχουμε τις ανταλλαγές απόψεων τις τροπολογίες ε, και θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Στη συζήτηση θα έχει σημασία η παρουσία σας. Τη μέρα που θα είναι η ψηφοφορία. Ίσως λιγότερο. Κύριε Γκουαλτιέρη. Εγώ αντικαθιστώ τον Σανφό Γιάννετς που είναι σκιώδης για την έκθεση αυτή. Απλώς θα εκφράσω κάποιες προτάσεις για τη γνωμοδότηση που εν γέρι μου φαίνεται καλή. Θα παρακαλέσω την εισηγητρία αν το θεωρεί σκόπιμο υπό το φως και ορισμένων παρατηρήσεων του συντονιστή για την ε, αντιμετώπιση της δημοκρατίας να δώσουμε μια πιο σαφή διατύπωση για ορισμένα στοιχεία, συστατικά θα έλεγα, της ε, αναφοράς στο ευρωπαϊκό πλέγμα για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Η εξωτερική διάσταση είναι πολύ σημαντική φυσικά. Και γι' αυτό θα ήθελα να ξανακοιτάξουμε λίγο την νομοδότηση, να την εμπλουτίσουμε θα έλεγα. Στη δε ανακοίνωση της Επιτροπής που παρουσιάζεται και της ε, υποεπιτροπής μας νομίζω θα ήταν χρήση, μέσα σε γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα καλό να έχουμε την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής, μια αναφορά. Κυρία Λούσινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Χάνκης. Δύο παρατηρήσεις μόνο. Πιστεύω καταρχάς ότι η γνωμοδότησή σας παραγνωρίζει πλήρως την μη στρατιωτική ε, φύσεως αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ξέρω ότι είμαι στην υποεπιτροπή αμήνης, αλλά ε, θα ήθελα η ε, καταπολέμηση των αιτίων που οδηγούν στην τρομοκρατία, τη φτώχεια δηλαδή κατά κύριο λόγο, να μην παραγνωριστεί, γιατί βλέπω ότι δεν καταγράφεται στο αρχικό κείμενο. Επίσης, μόνιμη ανάμεξη άλλων κρατών ε, για την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων ε, δεν θεωρείται σκόπιμη για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εδώ πρέπει να πω ότι ανησυχώ ιδιαιτέρως Για την ε, ζώνη του Σαχίλ νομίζω ότι δεν είναι οι στρατιωτικές λύσεις καταλληλότερες. Έχουμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση που χρειάζεται τελείως διαφορετικά και ιδιαίτερα μέτρα. Η περιοχή λοιπόν του Ζαχέλ δεν νομίζω ότι μπορεί να μπερδευτεί στο ίδιο κείμενο και στην εξισωθεί προ προς την τρομοκρατία με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Έχω επίσης ανησυχίες και αμφιβολίες ως προς την εξωτερική και εσωτερική διατύπωση μιας στρατηγικής που αναφέρεται στο κείμενο γιατί νομίζω ότι αυτό ισοδυναμεί με το να ανοίξουμε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο ρητά απορρίπτει η ομάδα μου. Αποτελεί τεράστια δε, τεράστιο δε κίνδυνο για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Κύριε Κόμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάνκης για την έκθεσή της. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά αυτά που μας είπε. Δίνει την προοπτική της υποεπιτροπής μας, συμπληρώνει τα όσα έχει η κυρία Ινετφέλτ περιλάβει στην έκθεσή της. Θεωρώ ότι αυτά που έχει πει η κυρία Ινετφέλτ δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε εμείς στην γνωμοδότηση, αλλά Ίσως να ήταν ε, καλό να επισημάνουμε κάπου ότι κανονικά εμείς ε, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με τα θέματα της ασφάλειας. Και θα έπρεπε επίσης εμείς να είμαστε εκείνοι που θα υπογραμμίσουμε ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία εάν ε, υπονομεύουμε τις δικές μας αξίες, δηλαδή αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με τον τρόπο αυτό παίζουμε το παιχνίδι των τρομοκρατών. Αυτό ακριβώς αποσκοπούν. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν. Το βλέπω στην έκθεση κυρία Σνετφέλτ, αλλά πιστεύω ότι δεν βλάπτει να πούμε και εμείς από πλευράς μας να επαναλάβουμε αυτές τις θέσεις. Και ιδιαίτερα όταν ξέρουμε πόσο σοβαρά είναι τα σφάλματα που έχουν υπό την πρόφαση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας οδηγήσει ουσιαστικά στην ενίσχυση των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα εκτιμώ την αναφορά στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το EFTP και άλλα σημαντικά προγράμματα. Ξέρω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υπεύθυνη παρακολούθηση της υλοποίησης ε, του προγράμματος συμφωνίας αυτής. Αλλά αυτό που χρειάζεται πιστεύω είναι εν γέννη να παρακολουθούμε την υλοποίηση όλων αυτών των συμβάσεων περί ε, κατά πολέμηση τη τρομοκρατία που έχουν επικυρώσει τα περισσότερα κράτη-μέλη. Όχι όλα, και αυτό βέβαια είναι λόγο ανησυχία, αλλά να κοιτάμε και πώ τι εφαρμόζουν. Έχω σοβαρέ τουλάχιστον αμφιβολίε για τι πρακτικέ που ακολουθούν ορισμένα κράτη-μέλη, περιλαμβανομένη και τη πατρίδα μου, ε, έναντι των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει. Και έχω και εμβολίε για το κατά πόσο είναι σοβαρή αυτή η προσπάθεια καταπολέμηση τρομοκρατία. Μέχρι ότου λοιπόν ε, καταπολεμήσουν ε, και ελέγξουν τις ε, υπεράκτιες εταιρείες όλες τις κυβερνήσεις δεν έχουμε κάνει τίποτα κατά της τρομοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μόνο κροϊδεύουμε τους πολίτες. Κατά την απόψη μου. Επίσης συμφωνώ με την κυρία Χάνκης εκεί όπου λέει ότι υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ και ανταλλαγή απόψεων και δράσεων μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των αντίστοιχων ε, δομών των κρατών. Το πρόβλημα που βλέπω πάνω απ' όλα είναι ότι υπάρχει μεταξύ των εθνικών κρατών κυρίως ανταγωνιστική σχέση και διάφορες ε, ε, υπηρεσίες μέσα στο κάθε κράτος, ε, άλλες στρατιωτικές δομές, άλλες πολιτικές δομές, διάφορες πολιτικές δομές μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Ε, πρόκειται για ένα χάος. Και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς προς κυβερνήσεις μας να πούμε ότι πρέπει πια να τα συγκυρίσουν όλα αυτά και να τα ελέγξουν. Ιδάλλως αποτελεσματικότητα δεν πρόκειται να υπάρξει στην καταπολέμηση τρομοκρατίας. αν δεν ε, συνεργάζονται μεταξύ τους εθνικές μας υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακόμη λιγότερο μάλιστα και σε εθνικό επίπεδο, δεν πρόκειται ποτέ να καταλήξουμε σε κάποιο σωστικό αποτέλεσμα. Και ξέρω ότι μιλάω περισσότερο έχοντας υπόψη την Πορτογαλία, αλλά είναι βέβαια ότι δεν είναι η μόνη ε, που, έχει αυτό, που δίνει αυτό το παράδειγμα στην Ευρώπη. Ο κύριος Πάσκου δεν ακούγεται. Ο κύριος Πάσκου χωρίς μικρόφωνο. It's Ναι, α προσπαθήσω να απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα, μήπω με καταλάβετε καλύτερα. Γιατί <laughs> και πιο σύντομη. Για την πρώτη ερώτηση. Ομολογώ ότι δεν την κατάλαβα εγώ αυτή τη φορά ω προ την εξωτερική διάσταση. Ε, τα 1600 χαρακτήρε που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω για τη γνωμοδότηση 1600 στοιχεία, με υποχρεώνουν να περιοριστήσω ένα πολύ στομό κείμενο. Ε, μέσα στο κείμενο όμω παρόλα αυτά βρίσκεται την εξωτερική διάσταση και ένα κατάλογο και των περιφερειών στι οποίε αναφέρομαι. Φυσικά είμαι διατεθειμένη το επεκτείνω περισσότερο, αλλά δεν μου επιτρέπεται περισσότερο χώρο. Αυτά λένε οι κανόνε. Επίση δεν κατάλαβα πολύ καλά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια παραπομπή, μια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Νετφέλτ, ένα έγγραφο το οποίο μάλλον δεν έχει πολύ μεγάλη επίδραση ε, ως προς τις πτυχές της δικής μας της αρμοδιότητας, γιατί αγγίζει άλλα θέματα. Άρα το μόνο πράγμα, το μόνο κείμενο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε αναφορά είναι ακριβώς η ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της δημοκρατίας εάν ε, δεν παραπέμπουμε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο έγγραφο, ουσιαστικά επαφίεται σε μένα να διατυπώσω ένα πρόγραμμα δράσης κατά της τρομοκρατίας, το οποίο βέβαια δεν είχε και πάρα πολύ νόημα. Εξωτερική δράση, εξωτερική διάσταση. Λέτε ότι την έχω λησμονήσει κυρία Λεωσίνη. Όχι, δεν νομίζω. Υπάρχει εσωτερική διάσταση, η εναρμόνιση της εσωτερικής με την εξωτερική. Τα αναφέρω όλα αυτά. Η ΔΕ Επιτροπή των Πολιτικών Υποθέσεων στην ε, έκθεσή της, ε, της κυρίας Σινετφέλτ δηλαδή, τα καλύπτει επίσης. Εγώ πολύ ευχαριστώ να αναλάβω να κάνω μια μακροσκελή έκθεση. Αλλά σε μια γνωμοδότηση μέσα δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτή την ε, ε, περιστασιακή αναφορά μόνο. Επίσης, για τα κονδύλια, ναι, ε, είναι αιτιολογημένη η παρατήρησή σας. Πλην όμως πρέπει να πω ότι ο κύριος Λόπες Ντεμπέλγκα νομίζω ήταν εκείνος ε, ο υπεύθυνο της δραστηριότητας ανάπτυξης αυτών των δράσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν γνωρίζω πολύ καλά το όνομά του, ίσως να το λέω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ε, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικά πράγματα και για λόγους προτεραιοτήτων ε, στην ανθρωπιστική δράση. Θα ήταν σκόπιμο να φτάσουμε στη ρίζα της ε, τρομοκρατίας, τη φτώχεια δηλαδή, και θα είναι καλό να το πούμε, αν και πολλέ φορέ μα λένε ότι δεν είναι καλό να μιλάμε τόσο περίφραστα μέσα σε γενικά κείμενα, σαν ένα κείμενο γνωμοδότηση δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συμφωνώ με την παρατήρηση σα και πολύ ευχαριστώ να την ενσωματώσω στο κείμενο. Κυρία Γκόμε, συμφωνώ με την πλειονότητα των παρατηρήσεών σας. Έχουμε άλλωστε συζητήσει τα θέματα αυτά όταν ε, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για το θέμα των ε, χημικών, βιολογικών και πυρηνικών απειλών. Ε, το θέμα που έχω ως πρόβλημα σε σχέση με την έκθεση Νετφέλτ και το βλέπουμε ως ε, κλασικό μοτίβο σε επίπεδο Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών είναι ότι έχουμε αφενός το μέλημα της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη και της ασφάλειας από την άλλη μεριά και αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ε, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί κάποια χρυσή τομή, μια ισορροπία ε, η οποία ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και διαφορετικά επιχειρήματα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μερικές φορές μιλούν μόνο υπέρ της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πολλές φορές για επικοινωνιακούς μονολόγους, ε, χωρίς να λαμβάνουν δηλαδή υπόψη το δικαίωμα του πολίτη, του ιδιώτη στην Ευρώπη να έχει ασφάλεια, να έχει επαρκή ασφάλεια, ασφάλεια επί την οποία εγώ κρίνω ως δικαίωμα εξίσου ε, θεμελιώδες, όσο και αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, έχω διατυπώσει 14 ερωτήματα προς την κυρία Ινετφέλτ, όπου τη ρωτώ πώς μπορεί το εγχείρημα το οποίο περιγράφει να υλοποιηθεί. Γιατί θα έπρεπε ουσιαστικά να μετατραπούν αυτά σε πράξη. Απάντηση δεν έχω λάβει όμως. Παράδειγμα, εκεί όπου γίνεται λόγος για έλεγχο του συνόλου των δαπανών, των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Να μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει όλο αυτό το θέμα στην επικουρικότητα. Είναι θέμα των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει, να επαληθεύσει, να μελετήσει εκ του σύνεγγυ τα στοιχεία τα σχετικά με του προπολογισμού, με τι δαπάνε των ημιστικών υπηρεσιών. Και ξέρω ότι στο Κοινοβούλιο δεν, έχω εγώ την, δεν εκφράζω εγώ την πλειοψηφία με τι θέσει αυτέ, αλλά εκφράζω τι δικέ μου θέσει, τελευταία τι προσωπικέ μου θέσει. Μετά, άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με κατάρτιση. και την ιδέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ε, βλέπω ότι η κυρία Νετφέλντ ουσιαστικά, επιμένοντας μόνο στα προσωπικά δεδομένα, υπονομεύει την ασφάλεια του πολίτη. Η δε συμφωνία που ανέφερε η κυρία Γκόμες στη FTP, ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να λησμονούμε όταν την αναφέρουμε και την ε, FNR, Μην ξεχνάμε όμως ότι όταν ήρθε η ώρα να συζητηθούν αυτά τα πράγματα, πολλοί βουλευτές ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες, στοιχεία, απάντηση όμως και συγκεκριμένος ορισμός για το τι είναι profiling και συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που δεν θα έπρεπε να δίνουν τέτοια στοιχεία, δεν είδα πουθενά. Ρωτώ λοιπόν εσείς πώς θα το χειριζόσταν το θέμα αυτό. Ομολογώ ότι δεν έχω καμία έτοιμη λύση, αλλά δεν είμαι και διατεθειμένη να αφήσω απεριόριστη πρόσβαση στον ιονδήποτε σε προσωπικά δεδομένα. Για τις υπεράκτιες εταιρείε και τους υπεράκτιους λογαριασμούς, βεβαίως πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα αυτό και να το συζητήσουμε. Η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ μυστικών υπηρεσιών είναι γνωστή, δεν έχουμε το χρόνο να την αναλύσουμε περισσότερο. Ξέρουμε πάντως ότι αυτή η ακριβώ ανταγωνιστική σχέση είναι που προξενεί δυσκολίε ω προ τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών είτε του ίδιου κράτου μέλους είτε γειτονικών κρατών μελών και ε, οδηγεί στα γνωστά προβλήματα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίω θα προσπαθήσω να ενσωματώσω τι προτάσει σα στο κείμενο στο βαθμό του δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Κατά θεστροπολογείο νέο στι 3 Μαου. Δεύτερη εξέταση 24 Μαΐου στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κλείνω το θέμα αυτό και τη συνεδρίαση προς το παρόν. Αύριο έχουμε ανταλλαγή απόψε μια σερβική αντιπροσωπεία βουλευτών για το θέμα της ασφάλειας πάλι. Είναι η μόνη δουλειά που έχουμε αύριο. 9.30 ξεκινάμε.